Okay. Okay, if you could uh, take your seats. Um. Καθίστε παρακαλώ. Χρειάζεται κάποια απαρτία για ορισμένα θέματα. Θα ξεκινήσω όμως με τις ανακοινώσεις του Προέδρου, της Προέδρου. Καλωσόρισα τα νέα μέλη μας από την Κροατία στο τέλος της συζήτησης για το νομισματικό διάλογο, χτες όταν ήταν και οι δύο παρόντες. Μετά την αφήξή τους ε, υπήρξε μια αλλαγή στο γλωσσικό καθεστώς. Έχω ήδη κάνει κάποιες ανακοινώσεις γύρω από αυτό Ξέρετε ότι ο κώδικας συμπεριφοράς για την πολυγλωσία είναι μια σειρά κανόνων που διέπουν την διερμηνία και τη μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία από τα, ένα από τα προαπαιτούμενα είναι ότι θα πρέπει να καθορίζει το, γλωσσικό της καθεστώς η ε, Επιτροπής μας επί τη βάση των πραγματικών αναγκών στην αρχή της εντολής και αυτό το αναλαμβάνει να το ελέγχει η Γραμματεία. Λαμβάνονται υπόψη λοιπόν και τα μέλη, τα τακτικά, και ανάλογα και με τις αίθουσες που έχουμε με διαφορετικό αριθμό α, α, <clears throat> θαλάμων κάθε φορά λόγω ακριβώς και των φυσικών αυτών περιορισμών μερικές φορές ορισμένες από τις γλώσσες τις συμπεφωνημένες θα έλεγα δεν είναι διαθέσιμες. Υπολογίζω στην κατανόησή σας γιατί δεν είναι δυνατό να έχουμε όλες τις αίθουσες εξοπλισμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες, τις 23 γλώσσες της Ένωσης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε ακριβώς τον αριθμό αυτό ανάλογα με το γλωσσικό μας προφίλ. Τώρα, οι τροπολογίες για τη γνωμοδότηση μετά από την υιοθέτηση του προϋπολογισμού για το 2014 από την Αυμόδια Επιτροπή. Η προθεσμία θα ξεκινήσει σύντομα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι θα πρέπει επίσης να αναφέρεστε στις τροπολογίες σας στο ποσό που ε, περιλαμβάνεται στην πρόταση προϋπολογισμού και όχι στη διαφορά την οποία θα επιφέρει η δική σας τροπολογία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η πρόταση του Συμβουλίου 5 Ιουλίου δεν ήταν διαθέσιμη. Η προθεσμία λοιπόν είναι η 18 Ιουλίου. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με τους αριθμούς να ζητήσετε πληροφορίες από τη γραμματεία μας. Η διαβούλευση της ΕΚΟΝ για την βελτίωση της συνεκτικότητας ε, είναι κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο πήραμε 86 απαντήσεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους απάντησαν και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για τον τριμερή διάλογο για το ΜΙΦΕΔ προβλέπεται να ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου σχετικά με την επιχειρηματική διακυβέρνηση θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και έχουν συμφωνηθεί και περαιτέρω τριμερείς διάλογοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται για τις 4 Σεπτεμβρίου. Okay. Oh. Okay. Right, Uh, we just, just uh, seem to have got a multiplicity of... Υπάρχουν διάφορα στο σημείο 7 Βασικά είμαστε στο επίπεδο της εκ νέου διαβούλευσης με την Επιτροπή στα πλαίσια του στατιστικού των στατιστικών επί τη βάση εν πάση περιπτώσει του άρθρου 70 του κανονισμού. Έχει ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει με τον Σικλούνα και ε, συνεχίζεται με τον Χουανγκόγκ Έχουμε ολοκληρώσει με μια γραπτή διαδικασία για το ευρωπαϊκό στατιστικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Θα ήθελαμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε μια νέα διαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει με κάποιο σχόλιο ή αν είμαστε ικανοποιημένοι από την διέξοδο των συναντήσεων και των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα που είναι πράγματι σαφές ότι υπήρξε αρκετή πρόοδος. Θα προβλεφθεί μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια, μάλλον στην Ολομέλεια του μηνός Οκτωβρίου. Η επόμενη εκ νέου διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά ε, <clears throat> ε, τις καταχρήσεις και χειραγωγήσεις της αγοράς πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Νομίζω ότι και εδώ στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος και θα δώσω σύντομα στην Άρλιν Μακάρθη το λόγο. Δεν θέλω να πω διάφορα ε, αλλά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική προσπάθεια την οποία έκαναν. Παρακολούθησαν από πάρα πολύ κοντά τα θέματα τα οποία ήταν ιδιαίτερο περίπλοκα και σύνθετα και να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της Γραμματείας και των πολιτικών ομάδων και της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής και το σύνολο του προσωπικού του Κοινοβουλίου που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας βοήθησαν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η πρόοδος προς την Αρλίν, σε ευχαριστώ για την αποτελεσματικότητά σου στα πλαίσια αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων. Μπορώ επίσημα λοιπόν επί τη βάση ε, των αποτελεσμάτων του τριμερούς διαλόγου να το συζητήσω μαζί σας εφόσον το επιθυμείτε ή εφόσον συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν τώρα για την απαρτία είμαστε 26 παρακαλώ μπορείτε να μετρήσετε τα μέλη. Λοιπόν, νομίζω ότι ίσως χρειαστούμε τις κάρτες μας για την ψηφοφορία, θα δείξει. Το θέμα είναι να ε, δούμε αν συμφωνούμε για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ε, τριμερούς διαλόγου. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την απόφαση αυτή λοιπόν, να αρχίσουμε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο βάσει του κειμένου που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και κυκλοφόρησε, ε, το έχει διανύμει η Γραμματεία, ε, με τη γνωστή διαπραγματευτική ομάδα, πρόεδρος, ε, εισηγητής και σκιώδης εισηγητές βασίζεται στο άρθρο 72 του κανονισμού η διαδικασία αυτή και θα πρέπει να εγκριθεί με πλειοψηφία ε, των μελών της Επιτροπής Οικονομικών όπως σας ανακοίνωσα χθες, είμαστε πλέον 50 τακτικά μέλη, αισίως με την έλευση των Κροατών συναδέλφων, οπότε η πλειοψηφία είναι 26 και θα πρέπει 26 να υπερψηφίσουν. Είναι η ψηφοφορία αυτή με βάση τον νέο κανονισμό. Υπέρ παρακαλώ τη έναρξη διαπραγματεύσεων τη εντολής δηλαδή. Okay. Anybody against? Μου κανείς κατά. Αποχή. Όχι. 29 υπέρ. 30. Χωρίς ε, αντίθετη ψήφο. Ευχαριστώ πολύ. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν λοιπόν. Τι περίπλοκα που είναι όλα αυτά. Ε, θα πρέπει να πάμε τώρα στο σημείο παρακαλώ 17 της ημερήσης διάταξης που είναι η ε, γνωμοδότηση της υποφαινομένης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Ε, βασικά τι έκανα εγώ εδώ. Προτάσεις βασιζόμενοι στην εμπειρία που είχαμε στην Επιτροπή μας στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Συγγνώμη, κάνετε πολύ φασαρία. I'll continue when it's quiet. Θα περιμένω να λίγο η αίθουσα για να συνεχίσω. Για να μπορώ να ακούω τη φωνή μου, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το πρώτο που θέλαμε να πούμε είναι ότι στον κανονισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουμε ε, τις τεχνικές πλέον ε, κανονιστικές προδιαγραφές και θέλουμε επίσης ε, όπου αυτό είναι δυνατό να εφαρμόζεται αντί των κατεξουδότηση πράξεων. Αυτό το συμφωνήσαμε στην υπόθεση μας σε Omnibus 1. Ε, και είναι ο σωστός ε, τρόπος κατά τη γνώμη μας να προχωρήσουμε. Επίσης θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δέχεται ε, τεχνική διαβούλευση από τους αρμοδίους για τις εγκατοξιοδότηση πράξης. Οι συνομοθέτες επίσης θα πρέπει να έχουν στόχο να δια διευκρινίσουν το πλαίσιο που εφαρμόζεται στο επίπεδο 1, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιλογές πολιτικής. Για παράδειγμα, ε, στο EFMD είχαμε μια εμπειρία αντίστοιχη χωρίς ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ΕΣΜΑ, πήγε στην καταξιοδότηση πράξη και τώρα όταν εμείς ε, έχουμε κείμενα επίπεδου 1 πρέπει να δίνουμε κατευθύνσεις, καθοδήγηση πολιτική και να είμαστε βέβαιοι ότι έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να γίνεται στην κανονική διαδικασία, να είναι ρουτίνα. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ο χρονικός ορίζοντας. Πολύ συχνά όταν προτείνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το διεκπεραιώνουμε εμείς μέχρι την τελική ψηφοφορία όσο γρήγορα θα επιθυμούσε ή θα φιλοδοξούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε σαφή εικόνα κάθε φορά του χρόνδιαγράμματος για ε, το ε, RTS και τις κατεξοδότηση πράξης. Για παράδειγμα σήμερα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που έχουμε ε, ακριβώς το πρόβλημα των εκλογών για ε, την αδηγία για τις κεφαλικές απαιτήσει. Αν είναι του χρόνου τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει κανείς. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε την πλήρη διαφάνεια όσο και τη διαβούλευση των ε, ενεχομένων σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και στο τέλος προτείνω και κάτι σε ένα σχόλιο για την ε, ίδια την ομάδα των ενδιαφερομένων, των ενεχομένων ε, θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι παρόντα σε αυτή την ομάδα των stakeholders δεν έχει να κάνει απαραίτητο με τις κατεξουδότηση πράξεις άμεσα, αλλά έχουν λόγο και γνώμη και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό να ληφθεί υπόψη και να λαμβάνεται γενικώ υπόψη. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ερμηνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Συμφωνία Πλαίσιο της Επιτροπής, ε, πράγμα που δυσκολεύει και βαραίνει τη διαδικασία και δεν μπορούν οι εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου κάθε φορά να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των ε, εμπειρογνωμόνων. Και πώς έχει η κατάσταση συχνά. Στη θεωρία ζητούν να στείλουμε επιστολή και να ζητούμε να παρευρισκόμαστε σε κάθε μία από τις συνεδριάσεις. Μα αυτή είναι ανέφικτη διαδικασία έχουμε μία ad hoc διαδικασία. Δεν μπορούμε σε κάθε φορά ε, να ζητούμε. Ζητούμε αναπερίπτωση, αλλά το ερμηνεύει με πάρα πολύ ατυχή τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχουν και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο από εμά να ε, βρεθούν σε ίση μοίρα και ίση μεταχείριση με τα κράτη-μέλη. Γιατί πολλέ φορέ ισχυρίζονται τα κράτη-μέλη ότι συζητούν θέματα στα οποία δεν επιτρέπεται εμεί να συμμετέχουμε, ενώ συζητούν και κατεξοδότηση πράξη και άλλα που μα αφορούν και πρέπει να συμμετέχουμε. Πρόσφατα ε, εγκρίθηκε ο κανονισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και ε, είδαμε και πάλι τα χρονοδιαγράμματα για τις τεχνικές κανονιστικές προδιαγραφές. Ε, ένας μήνας είναι ένα μήνα αν θυμάστε. Θα πρέπει επίσης να μην λησμονούμε το γεγονός ότι είναι συχνά περίπλοκα και ογκώδη τα θέματα αυτά και ουσιαστική η νομοθεσία. Εκεί λοιπόν τι κάναμε. Πήγαμε στο τρίμηνο, ένα συν ένα συν ένα. Ο τρίτος μήνας βέβαια είναι εφεδρεία και ε, θα μπορεί να χρησιμοποιείται όταν είναι αρκετά ογκώδης, αρκετά περίπλοκο το θέμα και ε, δυσκολίες σε σχέση με την ε, ολομέλεια και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί όταν πρόκειται να απορρίψουμε κάτι, η εμπειρία και πάλι έχει δείξει ότι χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο ανάμεσα στην ψηφοφορία, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε σε όλους περί τίνος πρόκειται για τα παράγωγα είχε επικρατήσει ένας πανικός. Είχαμε ε, ανησυχίες και θεμητές, αλλά οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θεώρησαν ότι ε, υποκύπταμε σε διάφορα λόμπι για την ομοθεσία, πράγμα που απέχει πόρο από την πραγματικότητα. Σε περίπτωση λοιπόν που ενδεχομένως να απορρίψουμε κάτι στην Ολομέλεια χρειαζόμαστε χρόνο είτε να εξηγήσουμε ε, την απόψή μας είτε να ε, αναζητήσουμε ένα συμβιβασμό. Και δεν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό προτείνω ένα μήνα συν ένα συν ένα, αν χρειαστεί. Και μάλιστα αυτό να είναι κανόνας. Επίσης, ασχολήθηκα και με το θέμα των θερινών διακοπών και για τις εκλογές θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην χαθεί όλος ο χρόνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, δώσει αρκετή ε, προσοχή σε αυτό και αρκετά νωρίς και μπορεί να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και το προγραμματισμό. Σε γενικές γραμμές αυτά είχα να σας πω. Είναι μερικά ακόμα αλλά εύκολα σε κατανόηση, δεν χρειάζονται εξηγήσει. Ε, αν είχατε καμιά δυσκολία στα εφαρμοστικά μέτρα στις κατεξοδότηση πράξης, παρακαλώ να μας το πείτε, να κάνετε και άλλες προτάσεις και τροπολογίες για να βελτιώσουμε το κείμενο. Τώρα δεν ξέρω. Αν έχουμε σκιώδεις ηγητές παρόντες μια στιγμή να σας δω. You were uh, the shadow. Ο Βέρνερ Λάγκεν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχεις σχόλια να κάνεις. Σε ποιο σημείο είμαστε, ρωτάει ο κύριος Λάγκεν. Στο 17. Κατ' εξοδότηση πράξης. Ή επειδή το έχω εγώ το θέμα, συμφωνεί σε όλα. Το 17, συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Εγώ κάνω μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, ε, υπό το φως μεταξύ άλλων των τεχνικών προδιαγραφών κτλ. Δεν έχω ιδέα, λέει ο κύριος Λάγκεν. Καλά beyond i think this is predominantly done from the chair δεν ξέρω μήπως θέλει κανεί το λόγο. Εδώ βασικά κυριαρχεί η πρόεδρος. Η Κέιτ και ο, η Κέιτ, Σουίμπον και ο Πέτερ. Ορίστε. Okay. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι σε σχέση με την γνωμοδότηση συμφωνούμε με την μεγάλη πλειοψηφία. Έχουμε μερικές προσθήκες, δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε τίποτα. Συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμα, με την ιδέα διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους, ε, τον νομικές σύμβουλες και την αξιολόγηση αντικτύπου. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτά τα μέτρα. Οι προσθήκες που θα ήθελα να προτείνω είναι για την ροή πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο και μέσα στην έκθεση μιλάτε ε, για πληροφορίες προς ε, το Προεδρείο και ε, στους εισηγητές. Θα έπρεπε επίσης να πληροφορούνται και οι σκιώδεις, διότι ό,τι προέρχεται από τους ενδιαφερόμενους, τους εμπλεκόμενους πρέπει να ενημερώνονται και οι σκιώδεις εισηγητές και θα είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε πλειοψηφία στην Ολομέλεια αν έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες εξ αρχής. Θα ήταν πολύ ευκολότερο αν αυτή οι κοινοποιήσεις επίσης γινόντουσαν προς τους κοιόδους. Έχουμε πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα για ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας μου θα ήθελα να προτείνω να ενσωματώσουμε μια ε, προφορική ανταλλαγή με την ΕΣΜΑ και για να μπορέσουν να καταλάβουν τα θέματα που απασχολούν το Κοινοβούλιο. Προτού όλα αυτά δημοσιοποιηθούν θα είναι εύκολο να διευκρινιστούν, εξηγηθούν ε, τα πράγματα ε, προτού δημοσιοποιηθούν. Αυτές είναι οι προσθήκες που θα ήθελα να προσθέσω, αλλά υποστηρίζω ε, το κείμενο. Περνάω στον Πίτερ. Ναι, και εγώ συμφωνώ Νομίζω ότι βεβαίως πρόκειται για τις δημοκρατικές αντιφάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εκεί όπου ένα επίπεδο, ε, ένα κείμενο ε, θα μπορούσε να απορριφθεί αν πάει προς μια κατεύθυνση την οποία δεν επιθυμούμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την κατανόηση, να το κατανοήσουμε αυτό ε, και αν αυτό περιληφθεί στο, σε όλη την διαδικασία με τη ΣΟΣΕΚΑ και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εργασία για την μεικτή επιτροπή επίσης και βεβαίως είναι κάτι εδώ στο οποίο, για το οποίο ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι η μεικτή επιτροπή όταν ε, τα εκπονήσουμε όλα αυτά να μας δείξει ε, πώς όλα αυτά προωθούν μια οριζόντια προσέγγιση και δεν το κάνουν και αυτό ε, θα πρέπει ε, να γίνει, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, μια τέτοια διαδικασία. Εγώ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ εφόσον έχω ορισμένα μέτρα, μέτρα εφαρμογής τα οποία πρότεινα. Ευχαριστώ, Σβέν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την εκθεσή σας, την οποία στηρίζουμε πλήρως. Πιστεύουμε ότι όταν πρόκειται για τα ίσας, ε, θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι η σύνθεση της ομάδας των ενδιαφερομένων για να μην υπάρξουν κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις ε, όταν θα ακολουθήσουμε την, τα μέτρα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα βασιστεί στις δικές μας διαδικασίες. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η πληθώρα των κατεξιοδότηση ε, πράξεων δεν έχουν πόρους, πόρους για μικρότερες ομάδες για να εργαστούν ε, με το προσωπικό που έχουμε εδώ, ε, για βοήθεια, για στήριξη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εργαστούμε πολύ δαλλιώσα θα είναι αδύνατον να κρίνουμε την ουσία όλων αυτών των πραγμάτων. Και επίσης έχουμε επίσης μια κατάσταση στην γραμματεία όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε όλα αυτά. Και όταν ε, θα έχουμε αποτελέσματα είτε από συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων είτε από, ε, σε σχέση με το, το νομοθετήματα δευτέρου επίπεδου ε, θα, θα υπάρχει ουσία που παρουσιάζεται αλλά δεν υπάρχει καμία κρίση, καμία αξιολόγηση διότι η γραμματεία δεν είναι ένα πολιτικό σώμα τουλάχιστον θεωρητικά. Συνεπώς αυτό ήταν αστείο βεβαίως που είπα. Και συνεπώς και συνεπώς υπάρχει το θέμα του πώς να καταστήσουμε εφικτή την ανάπτυξη ε, κρίσεων και εκτιμήσεων για τα διάφορα θέματα. Ε, δεν πρόκειται για μια κανονική νομοθετική διαδικασία. Υπάρχουν λίγες αιτήσει για σχόλια, για αλλαγέ. Όταν υπάρχουμε την κανονική διαδικασία υπάρχουν συνήθως πάρα πολλά σχόλια, ε, πάρα πολλές προτάσεις αλλαγών και τροποποίησεων. Ε, βεβαίως η Επιτροπή τα κάνει τα πάντα τέλεια, ίσως και τα διάφορα όργανα στο πρώτο μέρος της διαδικασίας. Αυτό είναι απίθανο βεβαίως. Συνεπώς υπάρχει ένα πρόβλημα νομίζω, ε, πρόβλημα ικανότητας να παρακολουθήσουμε, να δώσουμε μια συνέχεια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να προωθήσουμε, να προωθήσουμε, να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες σχετικά με το θέμα αυτό. Πολύ καλά. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Θα ήθελα απλώς... Ναι, ναι, ξέρω. Βεβαίως χαιρετίζω ε, το γεγονός ότι θα υπάρξουν προσθήκες. σύμφωνα με την ΚΕΙ ότι όλοι οι σκιώδεις ηγητές πρέπει να ενημερώνονται κατά κάποιο τρόπο ε, κυρίως σε μερικές περιπτώσεις που ζητούμε τυπικές επίσημες επιστολές. Ε, πόσο μπορούμε να ζητήσουμε να διαδίδονται, αν θα πρέπει να στέλνονται οι επιστολές αυτές σε όλους. Καμιά φορά είναι λίγο επικίνδυνο, δεν ξέρω ε, πού πρέπει να ε, απευθύνονται στο Προεδρείο, στην, ε, στις όταν βεβαίως η Πρόεδρος λαμβάνει αυτή την ενημέρωση, μπορεί να προωθήσει την ενημέρωση προς τον εισηγητή, αλλά αν προτείνεται μια τροπολογία, εγώ θα μπορούσα να κοινοποιήσω την πληροφορία αυτή σε πολύ περισσότερους. Πίτερ, νομίζω ότι ναι, θα ήταν καλή ιδέα να πούμε κάτι για τα οριζόντια θέματα και την μεικτή επιτροπή και ίσως επίσης είσαστε αυτός που έχει την μεγαλύτερη πείρα σχετικά με τα μέτρα εφαρμογή. και ίσως θα πρέπει να ελέγξουμε ότι έχουμε καλύψει αυτό το σκέλος δεόντος καταλήλως. Και σχετικά με την ομάδα των ενδιαφερομένων. Γι' αυτό ε, πρόσθεσα την, ε, το σημείο 9 ε, στο περιορισμένο χώρο που έχουμε σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε μετά να βάλουμε πολύ περισσότερα για την ομάδα των ενδιαφερομένων να συνδέσουμε με τα κατεξουσιοδότηση πράξεις Είναι σημαντικά όλα αυτά. Επίσης, πιστεύω ότι οι κανονικές, οι τακτικές ε, νομοθετικές ε, διαδικτασίες ε, επισύρουν περισσότερη προσοχή και το θέμα για με με τις πρότυπα τα ρυθμιστικά και τις πράξεις είναι ότι δεν επιφέρουν ουσιαστικά μέτρα πολιτικές. Εκεί ενσωματώνουμε αυτούς τους δείκτες πολιτικής όπου αυτή είναι απαραίτητη σχετικά με την νομοθετική διαδικασία. Αυτό που λείπει, που λείπει σε αυτήν την εντολή ε, λόγω ε, της πίεσης που έχουμε είναι ο χρόνος επιτροπής για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, συνέχεια παρακολούθησης διότι προσπαθούμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη και ελπίζουμε ότι στην επόμενη θητεία όταν θα έχουμε όλη τη νέα νομοθεσία για τις χρηματοπιστητικές υπηρεσίες και όταν περάσουμε στην επόμενη φάση θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για εξέλιξη εξέταση για έλεγχο δημοσίως επίσης. Αυτοί που ήμασταν εδώ στην προηγούμενη ε, θητεία ε, είδαν ότι μπορέσαμε να το κάνουμε με την οδηγία MIFID 1. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ε, διότι έχουμε λιγότερη πίεση και δεν έχουμε τόσες νέες πιέσεις. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής ε, που μπορώ να λάβω υπόψη όλα αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρατε ε, και αν θέλετε να μου στείλετε ένα σημείωμα αντί για τροπολογίες, πολύ καλά, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το, η προθεσμία είναι η 5η Σεπτεμβρίου στις 12 ε, και στις 23-24 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στις 30 ε, Σεπτεμβρίου πρωτού παραπεμφθεί. Για να δούμε τις αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι το 10 ε, το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίασης για τα μη πιστοτικά ιδρύματα εισήγηση πρωτοβουλία και την παρουσίαση από την εισηγήτρια την Κέι Σουίνμπερν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατανοώ ότι ε, το θέμα αυτό ίσως να μην ε, σας προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο πολύ όσο προκάλεσε το δικό μου και το δικό μου γραφείο. Το ενδιαφέρον είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα Λόγω ακριβώς όμως της φύσης του θα έλεγα, ακριβώς το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και η προσπάθεια ανάκαμψης είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα προσβλέποντας σε μελλοντικές κρίσεις γύρω από το θέμα αυτό. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι τα μη πιστοτικά ιδρύματα. Τα μη πιστοτικά ιδρύματα είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί και γι' αυτό είναι δύσκολο να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει τα πάντα. Εγώ θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε κρίσιμες υποδομές της αγοράς, τα ενδιάμεσα σώματα θα έλεγα, τα οποία ενσωματώνονται στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές και στα CSTs, όπου οι διαδικασίες αυτές ρύθμισης και διατησίας επιτρέπουν την ρύθμιση των προβλημάτων. Τα CCP και CSD λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη έκθεση. Έχουμε και άλλα πράγματα βέβαια τα οποία θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όπως την διαχείριση περιουσίας, ε, τις ασφάλειες λοιπά Είναι πάρα πολλά στον κατάλογο τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας και θα οδηγούμεθα στη συγκεκριμένη περίπτωση σε διεύρυνση ε, των ε, προβλημάτων, των αντικειμένων με τα οποία ασχολούμεθα. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται ένα επίσημο πλαίσιο για τέτοιου είδους κρίσιμες υποδομές. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια γενικότερη κρίση στην αγορά ή μια συγκεκριμένη επιχειρηματική κρίση, χρειάζεται να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ανεξάρτητα και διαφορετικά μάλλον από τις τράπεζες, όπου δεν μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο, είναι σαφές ότι εδώ θα επηρεαστούν και άλλου είδους δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές αρχές εκπροσώπησης έχουν κάνει σημαντικά βήματα σε σχέση με τον μηχανισμό ανάκαψης και εξυγίανσης. Νομίζω λοιπόν ότι η προσπάθεια της ε, CPSS αιοσκο είναι κάτι το οποίο έχει γίνει δεκτό και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει λάβει υπόψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της κρίσης της CPSS αιοσκο για τις επιμέρους χώρες έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα σε περίπτωση κρίσης. Ε, το θέμα της ανάκαμψης των τραπεζών, το οποίο ε, πέρασε και από τη δική μας Επιτροπή και από τον τριμερή διάλογο, δείχνει το πώς μπορεί να πτωχεύσουν οι τράπεζες εφόσον δεν είναι βιώσιμες. Όμως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποτύχουν και να πτωχεύσουν εκτός και αν αντικατασταθούν. Απαιτείται να υπάρχει μια ε, διαδικασία ανάκαμψης έτσι ώστε να συνεχίσουν αυτά τα μη πιστοτικά ιδρύματα να εργάζονται. Απαιτείται λοιπόν και το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις αυτές και εκτός του υπάρχοντος καθεστώτος φερεγγιότητας να λειτουργούν σωστά. Το θέμα είναι λοιπόν για τι χρειαζόμαστε, τη συγκεκριμένη δομή η οποία προτείνεται. Έχει μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσουμε ότι οι διαδικασίες ανάκαμψης είναι θα έλεγα το τεχνικό κομμάτι, το μη ένδοξο κομμάτι της διαδικασίας αυτής, αλλά επηρεάζει με συστημικό τρόπο την εσωτερική εθνική αγορά. Πρέπει λοιπόν ακόμα και οι μικρότερες τέτοιες επιχειρήσεις να διασφαλίζονται από διαδικασίες ανάκαμψης και εξυγίανσης και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι η συνέχεια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουν υπάρξει προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρξει ένα εναρμονισμένο καθεστώς ανάκαμψης και στις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν επί τη βάση του καθορισμού των αρχόδια βέρνησης να ε, καλύψουμε τις ανάγκες των CSTs. Ε, στην έκθεση μου προτείνω ότι όπου αυτό χρειάζεται οι επιχειρήσεις αυτές που λειτουργούν κάτω από πιστοτική άδεια θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρχές οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του πιστοτικού συστήματος, οπότε εφόσον χρειάζεται θα εφαρμόσουμε στις επιχειρήσεις αυτές το σύστημα που εφαρμόζουμε για την ανάκαμψη και εξυγίανση ε, των ε, πιστοτικών ιδρυμάτων. Θα υπάρχει βέβαια η δυνατότητα opt-out από το καθεστώς αυτός και αυτό και όχι η δυνατότητα επιλεκτικά opt-in στο καθεστώς αυτό και αναφέρομαι πάντα στα μη πιστοτικά ιδρύματα. Τα υπόλοιπα κρίσιμης φύσης CST, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός σε, κράτος, σε κάθε κράτος μέλος που θα επιτρέπει στην επιχείρηση αυτή να συνεχίζει τις δραστηριότητές της εκτός του ισχύοντος καθεστώτος Σε κάποιες χώρες αυτό γίνεται. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην πνίξουμε το σύστημα αν η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτύχει και περάσει σε καθεστώς έλλειψης φερεγγιότητας. Θα πρέπει οι λειτουργίες της να διασφαλιστούν, όμως με έκτακτες συνθήκες και κανόνες. Ε, αν είναι απαραίτητο μπορεί να δημιουργηθεί μια ε, υπηρεσία αν θέλετε ανάταξης ή ανάκαμψης που θα βοηθήσει ή θα μπορούσε η κεντρική τράπεζα να το αναλάβει αυτό έτσι ώστε να υπάρχει η νομική ασφάλεια που θα επιτρέψει τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Επί τη βάση των αρχών του CPSS IOSCO όλες οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται ασφαλιστικά. Έτσι, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την συνέχιση της λειτουργίας τους με έφετο τρόπο, σε έφετο χρόνο, συγγνώμη. Και αναφέρομαι στις υποδομές οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την αγορά. Ένα μεγάλο κομμάτι της υποδομής αυτής προέρχεται επίσης και ε, μετά από τις αναλήψεις υποχρεώσεων από πλευράς της ομάδας των 20. We now actually have a framework for the actual governance of σχετικά με τα CCP στην Ευρώπη και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τις βασικές αρχές ορθής διακυβέρνησης στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε τις δραστηριότητες αυτές για να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείρισή τους και έτσι θα πρέπει οι κυβερνητικές διαδικασίες να συνεισφέρουν στον περιορισμό των επιμολύνσεων που μπορεί να δημιουργηθούν στο εσωτερικό της αγοράς θα έλεγα να πούμε ότι τα μέλη αυτά έχουν σχέση με τα CCP ενώ δεν έχουν άμεσα οι επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να διασφαλίσουμε έτσι ώστε τα assets των πελατών να μπορούν να ελέγχονται επί τη βάση συγκεκριμένων εμπράκτων εγγυήσεων έτσι ώστε να καλύπτονται τα συμφέροντα ε, και της του ίδιου του CCP και των επιμέρους πελατών του. Ε, σαν παράδειγμα η κάλυψη, ο διαχωρισμός ορισμένων τέτοιου είδους περιουσιακών στοιχείων για τους πελάτες ε, ή θα πρέπει να διασφαλίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση η δυνατότητα μεταφοράς για να προστατευτεί ο πελάτης πρώτα και όλοι οι υπόλοιποι σε δεύτερη φάση. Απαιτείται λοιπόν σωστή διακυβέρνηση επιχειρηματική και ε, στην περίπτωση που υπάρξει αποτυχία ενός CCP ε, να υπάρχει ένα πλαίσιο ανάκαμψης ε, που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα της αγοράς και να λάβουμε υπόψη μας επίσης σαν κομβικό σημείο και την προστασία του επενδυτή. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα ταμείο αρκετά ισχυρό έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ε, των δύο μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην περίπτωση που αποτύχουν. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε, απίθανο στα πλαίσια της λειτουργίας της αγοράς να ζητήσει κανείς να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε έτσι ώστε το ότι η συνεισφορά των μελών να καλύπτει τις ανάγκες που θα χρειαστούν για την ανάκαμψη ε, των ευρωπαϊκών CCP. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί ε, ε, ακόμα και στην τελευταία κρίση να ξεπεραστούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών περισσότερο από τη συνεισφορά των μελών τους αλλά παρόλα αυτά η σημασία των CCP αυξάνεται και θα πρέπει να δούμε τι καθεστώτα θα πρέπει να δημιουργηθούν. Υπάρχουν περισσότερα προϊόντα τα οποία προσφέρονται και αλλάζουν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα, τα CCP, ιδιαίτερα σε σχέση ε, με τα θέματα της ε, διαχείρισης ε, των εμπράκτων εγγύησεων. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να εφαρμόσουμε τις αρχές CPSS ή OSCO. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πού σταματάει IOSCO. πού αρχίζει η διαδικασία, αν θέλετε, ε, πτώχευσης των επιχειρήσεων αυτών. Νομίζω ότι ε, εδώ είναι δύσκολο να βρούμε την διαφοροποίηση, το σημείο διαφοροποίησης. Προτείνεται στην έκθεσή μου ότι ε, ε, τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν στην περίπτωση όπου υπάρξει πιθανότητα πτώχευσης είναι μέτρα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες οι οποίες χρειάζονται. Αυτή στιγμή όμως έχουν τεθεί σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται τα έμπρακτα, οι έμπρακτες εγγυήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επιπλέον αρχή θα έλεγα η οποία να οδηγεί ε, στην CCP have failed. στην εξυγίανση της συγκεκριμένης, στην εκαθάριση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες γενικές απόψεις σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ συγκέντρωσα την προσοχή μου σε δύο τομείς τους οποίους έχουν υπάρξει υψηλή κίνδυνη στα CCPs και στα CSTs που έχουν συστημική σημασία και σε εσωτερικό επίπεδο της εθνικής αγοράς και σε επίπεδο ευρωπαϊκής αγοράς. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ένας μηχανισμός ανάκτησης αποτελεσματικός σε επίπεδο με τις παγκόσμιες βασικές αρχές της CPSS IOSCO. Το θέμα είναι πώς θα υπάρξει η δυνατότητα διαχωρισμού των διαδικασιών ανάκαμψης από τη μία και των διαδικασιών ρευστοποίησης από την άλλη. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα συμπεριλάβουμε και άλλους τομείς όπως τα συστήματα πληρωμών και επίσης ε, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κτλ. Νομίζω ότι οι αρχές CPISS IOSCO είναι ιδιαίτερα προχωρημένες σε σχέση με άλλους τομείς μη πιστοτικών ιδρυμάτων. Αν περιοριστούμε στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα επιχειρήσεων θα έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θέτουν προβλήματα διακυβέρνησης και τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία. Νομίζω ότι η αλληλοεπίδραση ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα έχει άμεση σχέση με την διακυβέρνηση των συγκεκριμένων μορφών επιχείρησης. Καλό θα είναι να μην αφήσουμε λοιπόν εκκρεμότητες και αυτό να γίνει με εύθετο τρόπο σε σχέση με την εμβέλεια. Ε, ξέρω ότι είναι πολύ τεχνικό, συγγνώμη που σας έκανα να βαρεθείτε, ε, εγώ θα ήθελα να και περιμένω με ενδιαφέρον τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ και να έρθουμε λοιπόν στους σκιώδεις. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η κυρία Ντανούτα Χούμπνε. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ. Επιτρέψτε μου να αρχίσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι αν θέλουμε σοβαρά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την υγιή λειτουργία των χρηματαγορών, θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε νομοθετικές κινήσεις, ε, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι τράπεζες. Ε, είναι σαφή τα λεγόμενα της και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη προς τα εκεί προσανατολίζεται για να εξηγιάνει το περιβάλλον λειτουργίας αυτών των Ιδρυμάτων και ενθαρρύνει ε, να γίνεται περισσότερη διακίνηση, ε, καθάριση λογαριασμών, διακανονισμοί κτλ. Ε, και θα πρέπει να δούμε και τα διάφορα εργαλεία που ανέφερε το ΕΜΙΡ, το MIFID κτλ. Ε, υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί που έχουν στόχο την πιο τακτική ε, λειτουργία την καθημερινή και χωρίς μεγάλους κινδύνους. Αλλά δεν καλύπτουν ε, έκτακτες περιπτώσεις και πάρα πολύ σοβαρές με μεγάλες πιέσεις και κραδασμούς. Χρειάζεται λοιπόν ακριβώς να ε, αναπτύξουμε σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης σε περίπτωση που διαταράσσεται η αγορά να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις. Και η έκθεση της ΚΕΙ πραγματικά μετατοπίζει τη συζήτηση προς την κατεύθυνση αυτή που θεωρώ σωστή. Επίσης η έκθεση εστιάζει σε ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την ε, εξυγίανση και ανάκαμψη ε, πιστοτικών ιδρυμάτων που δεν είναι τράπεζες. Μπήκε και σε πολλές λεπτομέρειες η συγγήτρια και θέλω να πω ότι το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε ορισμένα σημεία. Έχουμε το σχέδιο της έκθεσης και χρειάζονται ίσως μερικές συμπληρώσεις. Για τη γενική προσέγγιση θέλω πρώτα να πω το εξής για την ανάκαμψη και την εξυγίαση. Αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα, τα ίδια που δεν είναι τράπεζες, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αναπτύξουν τα ίδια ε, συνολικά προγράμματα τα οποία θα αναθεωρούν ε, η αρμόδια αρχή εμπροκειμένου και θα μπορεί να ζητά και αλλαγές σε αυτά τα σχέδια. Η εποπτική αρχή επίσης θα πρέπει να έχει την εξουσία να επεμβαίνει ε, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζει η αρχή ότι υπάρχει κίνδυνος να επέλθει ανασφάλεια και αβεβαιότητα στην αγορά, ιδιαίτερα υπό συνθήκες πίεσης. Αυτό το θέμα της εξυγίανσης ή της ε, καθάρισης ε, θεωρώ χρήσιμο να προσθέσουμε εδώ ότι οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να προσπαθούν να συνεργάζονται και να ενημερώνουν η μία την άλλη. Γιατί υπάρχουν όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, σε διάφορες δικαιοδοσίες και όταν πρέπει να εξηγιανθούν χρειάζεται συνεργασία όλων αυτών των αρμοδίων αρχών ε, στα διάφορα κράτη. Μπορώ να φανταστώ μια κατάσταση. Ε, που να ε, συγκρούεται με κάποιες εθνικές σκέψεις, αλλά θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι οποιασδήποτε μελλοντικέ ρυθμίσεις που θα διέπουν αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα θα πρέπει να συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία. Ξέρω, συμφωνώ και η σε αυτό. Επίσης πιστεύω ότι η ειδική φύση των κεντρικών αποθετηρίων αξιών χρειάζεται ε, ε, έναν ορισμό για τη λειτουργία τους. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί αυτός. Και στο σημείο 12 νομίζω η έκθεση πολύ σωστά αναφέρει ότι στο σενάριο κρίσης η βασική ε, λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων θα πρέπει να διασφαλίζεται και να είναι δεδομένη και να Υπάρχουν όμως και άλλες λειτουργίες καταγραφής ε, των ε, τίτλων και μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος ε, στο διακανονισμό. Δηλαδή, τι εννοώ, ε, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων έχουν ε, διάφορες λειτουργίες, ε, λειτουργία φύλαξης, λειτουργία καταγραφής. Ζητώ συγγνώμη, διότι απεχθάνομαι αυτά τα αρχικά και ακτικόλεξα και μπερδεύομαι. Ίσως μακρηγορώ γιατί δεν χρησιμοποιώ αρχικά, λέγω κεντρικά αποθετήρια τίτλων και όχι κάτ. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ε, το ρόλο των CCP, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων που έχουν άδεια ε, λειτουργίας ως τράπεζες. Υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς εκεί που χρειάζεται και ε, όχι το καθεστώς εξυγίανσης μετά την ανάκαψη των τραπεζών στην αντίστοιχη οδηγία. Εδώ έχω μια ιδιαίτερη ανησυχία. Το σύστημα που προτείνεται για τις τράπεζες απαιτεί ε, να συσσωρεύουν ένα χρέος το οποίο μπορεί να σώζεται ε, από μέσα, το bail-in δηλαδή. Αυτό είναι λίγο προβληματικό ε, γιατί συνήθως δεν εκδίδουν τέτοιους τίτλους χρέους. Και τέλος για τα συστήματα πληρωμών νομίζω ότι και εκεί χρειάζεται ένα σωστό σύστημα ανάκαμψης και εξυγίασης διότι απλούστατα είναι ε, στο κέντρο όλων ε, των ε, μεταφορών και με μετρητών ρευστών. Και αυτό μπορεί να επιμολύνει, να μετατεθεί σε άλλους φορείς της χρηματαγοράς. Αν δείτε τον διακανονισμό του 1999, την οδηγία δηλαδή, στόχο έχει να μετριάσει, να περιορίσει τους κινδύνους των συστημάτων πληρωμών, αλλά η οδηγία αυτή δεν καλύπτει επαρκώς ε, το πεδίο της ανάκαμψης και της εξυγίασης και χρειάζονται και διευκρινήσεις, ειδικέ ε, ρυθμίσεις γι' αυτό και ένα τελευταίο για τις ασφάλειες. Ασφαλιστικές εταιρείες στη σημερινή ε, εκδοχή ε, η ΚΕΙ απλώς το θίγει, δεν ε, επεκτείνεται σε αυτό. Ξέρω βεβαίως αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το γεγονός ότι πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις διάφορες εξελίξεις στο θέμα της φερεγγιότητας 2. Γνωρίζω την κατάσταση, έχει καθυστερήσει αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω πώς μπορούμε ε, να το εντάξουμε αυτό στην έκθεση της ΚΕΙ. Γενικά Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία στο παρόν στάδιο να κάνουμε αυτή την έκθεση. Η Case Swinburne έχει εργαστεί πάρα πολύ και ελπίζω αυτά που θα προτείνει και μαζί με τους σκιώδεις να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουμε λίγο να επηρεάσουμε τις προτάσεις της για αυτό το θέμα. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τώρα ο Λεωνάρντο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Σρίμπορν. E ε, Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο τεχνικά και ελπίζω και εγώ όπως και η κυρία Χούπνερ σαν σκιώδης εισηγητές να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με επικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον καθορισμό του νομικού και διακανονιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα επιτρέψει την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο και παρουσιάζει πάρα πολλούς κινδύνους και αναφέρομαι στην λειτουργία των κρισίμων υποδομών της αγοράς. Από την άλλη, ήδη με την προσπάθεια που έχει γίνει μέσω του κανονισμού ΕΜΙΡ, κάποιες προϋποθέσεις έχουν ήδη τεθεί επί τη βάση ακριβώς των νέων προτάσεων, αλλά το ΕΜΙΡ από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συνολικού πλαισίου παρεμβάσεων ε, σχετικά με την ε, επίλυση και την ε, εξυγίανση των σε κρίση επιχειρήσεων. Εγώ θα προσπαθήσω λοιπόν από πλευρά μου να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις και στα πλαίσια αυτής της πρώτης παρουσίασης θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και να εκφράσω κάποιες αξιολογήσεις σχετικές με αυτά τα οποία έλεγε η Κέι Σουίνμπορν. Ε, πριν από οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι αναμφίβολα υπάρχει ανάγκη να υπογραμμίσουμε την διαφοροποίηση, την πιο ξεκάθαρη διαφοροποίηση ε, των τμήματων που συναποτελούν την εμβέλεια της έκθεσης και ε, της συνολικής πρότασης που θα κληθούμε να, να υιοθετήσουμε. Θα συμφωνήσω με τη Σουίμπορν ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στα κεντρικά CCP και στους κεντρικούς καταθέτες και εδώ θα ήθελα να ε, κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Όμως δεν μπορούμε να αποκρύψουμε το ότι πολλά άλλα υποκείμενα τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια της αγοράς όπως τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων λόγω ακριβώς των ιδίων χαρακτηριστικών τους, της εμβέλειάς τους και της λειτουργικότητάς τους μπορούν να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερη μεγάλη συστημική σημασία, μεγάλο συστημικό βάρος και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι ε, έχουν άμεση σχέση με τα συστήματα της, τα, τα πιστοτικά όπως λέγονται και ε, εδώ να εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν και για τις τράπεζες σε σχέση με τη ρευστότητά τους και τα λοιπά. Νομίζω πάντως ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει να ανοίξει κάποια περιθώρια, να αφήσει συγγνώμη κάποια περιθώρια τα οποία ανακαλύπτουν όλους τους τομείς και τομείς οι οποίοι ε, αφορούν άλλου είδους κρίσιμες υποδομές αν και πάντα το κέντρο της ενασχόλησής μας είναι τα δύο θέματα στα οποία προαναφέρθηκα. Και να αναφερθώ εδώ κυρίως στο θέμα των ε, CCP's. Νομίζω ότι ιδιαίτερα μετά από αυτά τα οποία έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΕΜΙΡ για τις υποδομές της αγοράς, πέρα από αυτά που έχουμε κάνει λοιπόν μέσω του ΕΜΙΡ, ο ρόλος και η συστημική σημασία των CCP γίνεται κάτι το ακόμα πιο σημαντικό. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαρα τα προβλήματα τα οποία χαρακτηρίζουν την, ε, τις διαδικασίες ανάκαψης και εξυγίανσης. Το πρώτο θέμα το οποίο τίθεται είναι ότι σύμφωνα με τη δική μου άποψη θα πρέπει να δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι διαστάσεις και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των CCP. Είναι προφανές ότι ανάλογα με τον ρόλο και την διάσταση την οποία έχουν καθορίζεται και η συστημική τους βαρύτητα. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε ότι όταν ένα εθνικό CCP μπορεί να συνεισφέρει στην χρηματοδοτική σταθερότητα, τότε θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με τον ρόλο τον οποίο μπορεί να έχει ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εθνική Αρχή Εποπτείας. Έχω την αίσθηση ότι εδώ έχουμε ένα πρώτο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε σχετικά με την διαφοροποίηση ποιοτικά και την διαφοροποίηση ανάλογα με την εμβέλεια των συγκεκριμένων εθνικών CCP πάντα σε σχέση με τα CCP δεν θα ήθελα να μπω στις, να περάσω στις τεχνικές λεπτομέρειες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι αν και ε, υποτίθεται ότι οι αντισυμβαλόμενοι πρέπει να είναι πάντα σε ε, θέση να συγκεντρώσουν ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία συγκεκριμένη υπόθεση σχετικά με τους λεγόμενους χρήστες Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει μεγάλη σημασία γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα της συστημικής ισορροπίας λειτουργίας του συστήματος. Αλλά από την άλλη έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των χρηστών των αντισυμβαλωμένων των κεντρικών είτε με άμεσο τρόπο με αριθμό μέλους κατά κάποιο τρόπο ε, και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι η ξεκάθαρη η ε, επιθυμία μας να προστατεύσουμε αυτού του είδους τους χρήστες. Εδώ τίθεται ένα πιο γενικό ε, θα έλεγα ευαίσθητο όμως ταυτόχρονα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Το θέμα αυτό αφορά την δευτερογενή αγορά όταν δεν έχουν υπάρξει ε, διαπραγματεύσεις σε επίπεδο εγκεκριμένων διαδικασιών έτσι ώστε να αποφύγουμε χειραγωγήσεις και καταχρήσεις. Νομίζω ότι στα πλαίσια ε, της προσπάθειας της επίλυσης μιας κρίσης των αντισυμβαλωμένων θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες, πελάτες θα πρέπει να προστατεύονται και δεν θα πρέπει να ρίξουμε επάνω τους το πλήρες βάρος το οποίο θα προκαλέσει μια κρίση ή μια συγκεκριμένη δυσκολία. Για να κλείσω θα ήθελα να κάνω μία φορά ε, στους ε, CCPs οι οποίοι σαν πρότυπο θα έλεγα λειτουργίας δεν καλύπτονται από τις διαδικασίες εξυγίανσης και οι διαδικασίες ε, εξυγίανσης δεν είναι σε θέση να κεφαλαιοποιήσουν μια χρηματοδοτική ε, διαδικασία. Θα πρέπει να προβλέψουμε εδώ μια σημαντική λειτουργία των εποπτικών αρχών έτσι ώστε σε περίπτωση κρίσης να διασφαλιστεί η λειτουργική συνέχεια του συστήματος με τους κατάλληλους κάθε φορά τρόπους ακόμα και αν οι αντισυμβαλόμενοι έχουν χτυπηθεί από μια σοβαρή κρίση και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει έτσι ώστε να αποφύγουμε τις επιμολύνσεις και να διασφαλίσουμε ε, την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνέχεια. Αυτές είναι κάποιες πρώτες γενικές παρατηρήσεις. Παρ' όλα αυτά είμαι στην διάθεση της εισηγήτριας για να εμβαθύνουμε στο θέμα και για να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε πιο σωστά σε ένα θέμα πάρα πολύ τεχνικό και πάρα πολύ περίπλοκο, αλλά μέσα στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καινοτόμο και όταν επιδιώκει κανείς την καινοτομία οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Uh, thank you very much. Um, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης από πλευρά Άλντε. Γι' αυτό και θα μιλήσω τώρα. Σε ευχαριστώ και για την έκθεσή σου και για τα διαγράμματα στην αιτιολογική σου έκθεση. Ε, γιατί είναι όλο και πιο περίπλοκα τα θέματα και προσπαθούμε να τα καταλάβουμε. Για το πεδίο εφαρμογής το έθεσες και εσύ. Είναι δύο τα μέρη της έκθεσης ας πούμε. Το ένα είναι η κρίσιμη υποδομή και μπαίνει και σε λεπτομέρειες και πραγματικά εκεί ε, χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, απαντήσεις, παύλα, υποδείξεις, ε, προτάσεις για να συμβάλλουμε σημαντικά στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πρέπει να μας προτείνουν νομοθεσία. Και ένα δεύτερο μέρος, και το ανέφερες και εσύ, είναι κάτι που χρειάζεται να συνεχίσουμε να ερευνούμε. Ε, με αυτό το διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το ε, προτείνουμε και υπάρχουν προβλήματα ε, με την τίτλοποίηση και την κεφαλαιοποίηση, το skin in the game και πώς όλα αυτά συμβιβάζονται και συνδυάζονται. Αυτή τη στιγμή όλο και περισσότεροι επενδυτές ε, ζητούν να έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων τους και μπορεί αυτό να έχει επιπτώσεις ε, στην εκαθάριση ε, και στην πτώχευση και για την κρίσιμη υποδομή είναι επίσης κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ο Πίτερ θέλει να, κάτι να πει, τον έχω σημειώσει για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, αλλά και πάλι έχουμε μετατοπίσει λίγο τα προβλήματα των τραπεζών και ε, της ε, ανάκαμψης και εξυγίανσης προς τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι αυτοί θα υποστούν τη διάσωση, το bail-in δηλαδή, και δεν ε, υπάρχει ακόμα ρύθμιση για το τι θα ισχύσει για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιδοτικά ταμεία. Και το θέμα δεν είναι να πάρουμε μια κρίση και να μεταμοσχεύσουμε σε έναν άλλο κλάδο ε, των χρηματοπιστωτικών. Είναι ίσως πολύ νωρίς από τώρα ε, για να λύσουμε όλα τα θέματα, αλλά τουλάχιστον να τα επισημάνουμε. Από τις τράπεζες ε, μάθαμε πολλά όταν οι δύο πολύ μεγάλες τράπεζες που ήταν πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν προχώρησαν στα σχέδια ανάκαψης και εξυγίασης. Θυμάστε οι δύο too big to fail και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και προγραμματισμός. Ε, εγώ προσπάθησα αυτό ε, να το συμπεριλάβω στην νομοθεσία, το θέμα της ανάκαμψης και της εξυγίασης ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάτι άλλο. Ορισμένοι θα απευθυνθούν στις κεντρικές τράπεζες, πολύ μεγάλα συστήματα, γιατί ε, ε, για τα συστήματα πληρωμών, ας πούμε, έχουν οι κεντρικές τράπεζες λόγο και ρόλο ε, και είναι ένα από τα σημαντικά κεντρικά στοιχεία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα σημαντικότερα και μετά τι θα γίνει με τα υπόλοιπα όσα ε, χρειαστεί να προχωρήσουν σε κάποιες διαδικασίες να είναι ε, τακτικές και συντεταγμένες και όχι άτακτες. Να μην εγκλωβιστούν κάπου σε μια ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιος κατέχει, τι, ε, ποιο είναι το περιουσιακό στοιχείο καθενός, ε, τι χάνεται και τι διασώζεται. Καμιά φορά όταν ανασταλούν κάποιες απαιτήσει ε, μπορούμε να σώσουμε μια κατηγορία που είναι εγκλωβισμένη στο τράζιτ, στην ενδιάμεση αυτή η κατάσταση. Και Χαίρομαι που κάνεις προτάσεις για το κεντρικό αντισυμβαλόμενο, το CCP, που θα πρέπει να είναι ενδεχομένω στο όριο μεταξύ ανάκαμψης και εξυγίανσης, εκαθάρισης. και δεν ξέρω αν υπάρχει ας πούμε προτίμηση σε πελάτες ή προτίμηση καταθέτες για να πούμε ότι αυτός θα την πληρώσει τελευταίος. Ποιος? και καμιά φορά αυτός που θα την πληρώσει τελευταίος την πληρώνει, ε, αλλά άλλες φορές γλιτώνει. Και αυτά θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε, ε, να δούμε μέχρι πού θα υπάρξει ο παραλυσμός με τις τράπεζες. Τελικά οι καταθέτες χάνουν τα λεφτά τους. Βέβαια, όταν είναι ασφαλισμένοι, ε, μπαίνει η ασφαλιστική εταιρεία και τους πληρώνει. Άρα ρίσκο έχουν όλοι. Αυτό τι σημαίνει κάποιος που είναι πελάτης και έχει μπει σε μια δραστηριότητα αγοράς και ε, πώλησης παραγόγων. Θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί εξίσου να χάσει. Δηλαδή όταν έχει τα χρήματά σου σε μια τράπεζα και η τράπεζα καταρρεύσει μπορεί και να τα χάσεις, ακόμα και να είναι καταθέσεις. Αυτό θα πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να το καταλαβαίνει και να το αντιμετωπίζει. Άρα ε, δεν πειράζει να μειωθεί και λίγο η αγορά των παραγόγων. Επίσης ε, μιλάς για τους πελάτες ε, και την έμεση εκαθάριση για μικρές τράπεζες με τους CCP, τους κεντρικούς αντισαβαλωμένους. Αυτό είναι ε, μια ελαφρώς διαφορετική κατηγορία πελατών. Είναι πολύ σημαντική λειτουργία και δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτή. Είναι και πάλι μια ενδιάμεση κατάσταση. Εχθές ε, το συζητήσαμε στη συνεδρίαση που είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΕΜΙΡ, τον κανονισμό για τις υποδομές ε, των αγορών και τι γίνεται με τις υποθήκες ε, των εμπράκτων εγγύησεων και τι μπορεί κανείς να δεχτεί και τι δεν μπορεί να δεχτεί εκεί στις υποδομές. Πάντως, θα πρέπει οπωσδήποτε να γράψουμε στην έκθεση ότι η ΕΣΑ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ε, θα πρέπει να έχει ένα ρόλο συντονιστικό, να κοιτάει αυτά τα ζητήματα ανάκαμψης και εξυγίανσης και τα σχέδια. Αυτό το είχαμε και στον κανονισμό του EBA της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, αλλά τελικά χάθηκε. Ε, υπάρχει κάπου εκεί μια ε, εντολή στο κανονισμό 4 για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις, το CRD4, για να υπάρχει και ρύθμιση, ακριβώς γιατί αυτές οι δραστηριότητες είναι κατεξοχήν διασυνοριακές και μπορεί να έχουν και αντίστοιχες επιπτώσεις. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς και να παρακολουθούμε και τη διαδικασία και το διεθνές γίγνεσθε. Ε, έρχομαι τώρα στο CSD, φεύγω από το CCP στους κεντρικούς αντι, ε, συμβαλωμένους Τώρα, αν είτε είναι τράπεζε, είτε δεν είναι ορισμός ε, του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο κανονισμό για τις κεφαλαιτικέ απαιτήσει είναι ότι θα πρέπει να δέχεται καταθέσεις. Ε, υπάρχει και περιορισμός της άδειες και αυτό θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει και τι αντίκτυπο ή μπορεί και να μην επηρεαστούν καθόλου από το ε, σύστημα και την οδηγία για την εκαθάριση εξηγίας των τραπεζών. Αν η διαφορά λοιπόν είναι οι καταθέσεις, ε, ε, μπορούμε έτσι να ρυθμίσουμε τι εμπίπτει σε ποια κατηγορία και τι όχι. Το ξεκαθάρισε και η Ντανούτα ότι υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της ενημέρωσης και επανέρχομαι ε, και στις υποθήκες θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ε, ποιος κατέχει τι, ε, πότε και πώς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η διαδικασία καταχώρηση κάπου καταγραφής να ξέρουμε όταν χρησιμοποιούνται εγγύησεις, εμπράγματες ευχαριστώ για την έκθεσή σου. Θα τη μελετήσω ε, ενδελεχέστατα το καλοκαίρι. Ε, ελπίζω να βοηθήσουμε να ε, περάσουμε σε κάποιους ορισμούς και να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Ελπίζω να βοηθήσουμε λοιπόν να προχωρήσει η έκθεση. Αυτά από τους φιλελευθέρους. Βασικά ήταν πολλά προσωπικά από τους πρασίνους, ο Ζαν Πολ. Ποιος θέλει, ο Μπάς Εκχάουτ. Ωραία. Λάθος είχα σημειώσει. Uh, Πολύ καλά, ναι. Πρώτα Άρχισα βεβαίως να ανησυχώ για τις καλοκαιρινές σας ε, διακοπές. Αν πρόκειται να τις περάσετε μελετώντας αυτό το κείμενο, ε, βεβαίω, ο Φιλίπ ε, Λαμπέρ ψηφίζει στην Ήτρα, είναι σκιώδη, αλλά θα προσπαθήσω ε, να αναφέρω τη δική του τοποθέτηση. Βεβαίω πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ τεχνικό. Αν πρέπει κανείς να αντικαθιστά τον σκιώδη, γίνεται πιο τεχνικά το θέμα για το άτομο αυτό. Από τη δική μα προοπτική, αν εξετάσετε πού είναι η εστίαση και βεβαίω ευχαριστώ πολύ όλες οι συστάσεις για τα CCP και τα CDS, όλα αυτά ε, βεβαίως ε, τα δεχόμαστε. Δεν βλέπω πολλά σημεία τα οποία θα θέλαμε να προσθέσουμε. Ε, θα ήθελα όμως να αναφερθώ εκεί όπου πρέπει να γίνουν προσθήκες κατά τη δική μας προοπτική. Σύμφωνα με μας πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τους ασφαλιστές και εμείς πιστεύουμε ότι αν εξετάστε ε, τι συνέβη με την ε, AIG ε, παγκοσμίως όταν υπήρξε η κρίση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποδώσουμε περισσότερη προσοχή για στους ασφαλιστές σχετικά με το θέμα της ανακάμψης και εξυγίανσης. Αναπιστεύουμε ότι εκεί όπου οι ασφαλιστές έχουν διασυνορικές δραστηριότητες και underwriting που σχετίζονται βεβαίως με ορισμένες ορισμένα μέσα, χρηματοπιστωτικά και προϊόντα επενδυτικά, νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ειδική, ειδική εξυγίανση για αυτή, για αυτή την κατηγορία. Αλλά νομίζουμε ότι όταν υπάρχουν διασυνοριακές δραστηριότητες πρέπει να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο σύστημα. Σχετικά με το σύστημα πληρωμών ε, και τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και στοιχείων ενεργητικού νομίζουμε ότι είναι πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα, πολλές, μη, πάρα πολλά μη πιστοτικά ιδρύματα που ασχολούνται με την, με την τιτλοποίηση και τέτοιες αγορές και υπάρχουν ε, συνέπειες για το χρηματοοικονομικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτά τα σώματα και πώς θα υπάρξει η παρακολούθηση και ίσως να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς εξυγίανσης. Αλλά πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε ε, τα, τους ενδιαφερόμενους τρίτο και τελευταίο σημείο που θα θέλαμε να επισημάνουμε, ήδη αναφέρατε ότι εκτός από την παρακολούθηση των κινδύνων επιμόλυνσης από ορισμένε τράπεζες σε αντισυμβαλόμενα μέρη, σε CCP, νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου θα έπρεπε να έχει ένα σύστημα παρακολούθησης του κινδύνου δικτύου λόγω της αλληλεπίδρωσης ανάμεσα σε πολλές χρήματο αλληλεπίδραση μεταξύ χρηματοπιστικών ιδρυμάτων και άλλων πρωταγωνιστών της αγοράς. Ίσως θα πρέπει να έχουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε την έκθεση αλλά όλες οι ε, συστάσεις για τα CCP και CDSD είναι ευπρόσδεκτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να λάβει τον λόγο. Όχι, αυτή τη φορά δεν έχω σχόλια πολύ καλά. Ο Πίτερ επίσης θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε το θέμα της AIG ε, που ήταν ένα σημείο σημαντικό αυτής της κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει δικαιολογία ε, μια τέτοια επιχείρηση να έχει με λόγω της ιδιοκτησίας της τέτοιες μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Διαρωτώ με εάν δεν θα πρέπει να προσθέσουμε περισσότερα στρώματα. Ε, βεβαίως ε, θα έχουμε μια απλή συζήτηση και όχι ε, πολύ περίπλοκη για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την κρίση μας για το τι πρέπει να γίνει. Ανησυχώ για τις συνέπειες για τους γενικούς ασφαλιστές σε σχέση με τους ασφαλιστές τραπεζών. Υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στην γενική τραπεζική και τις ασφάλειες υπάρχει κάποια ε, σύγχυση διότι ορισμένες ε, τράπεζες, πώς αντιμετωπίζουν οι τράπεζες ε, το δικό τους ισολογισμό και τους άλλους που πολλούν προϊόντα εντός εισαγωγικών μακροπρόθεσμα. Υπάρχει μια σύγχυση. Η Ντανούτα ανέφερε βεβαίω ότι όλοι θέλουν να ξέρουν πού βρισκόμαστε ως προς την φερεγγιότητα δύο και οι συνέπειες από ό,τι ακούμε και από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευρεπής λύση για μακροπρόθεσμη εγγύηση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία. Και είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε κάτι τέτοιο στη συζήτηση όσο θα αναπτύσσεται ο τριμερής ε, διάλογος και όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο που το Κοινοβούλιο θα έχει ε, κάποια συνένεση σχετικά με την ψηφοφορία. Αλλά νομίζω ότι ο τομέας των ασφαλιών είναι εξαιρετικά σημαντικός διότι εκεί το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων είναι μεγάλο αλλά η κίνδυνη είναι διαφορετική όπως είναι και η δραστηριότητα. Ε, επικροτώ τα όσα είπε η ΚΕΙ σχετικά με τις διεθνείς αρχές, κυρίως της AIAS, για να έχουμε ε, τις αρχές αυτές, αλλά να μην ε, ξεχνάμε το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Έχουμε τον διαχωρισμό ε, των στοιχείων του ενεργητικού, κάτι που δεν κάνουμε μέσα στο Κοινοβούλιο, να διαχωρίσουμε τις δραστηριότητες, την δίκηση από τα κονδύλια των επενδυτών. Ίσως θα πρέπει σε κάποιο σημείο να επανέλθουμε εδώ ε, και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε την κοινότητα των επενδυτών. Είναι κάτι που καλύψαμε σε προηγούμενη συζήτηση μέσα στην Επιτροπή Ε, μην, ε, και μην θεωρείς ε, ότι το λέω αυτό εχθρικά. Κάθε φορά όμως χρησιμοποιούμε τη σύγκριση με τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν ήταν πάρα πολύ επιτυχημένες δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ως αποτέλεσμα ίσως να πληρώνουμε άλλα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι στην αγορά ε, με τον ίδιο τρόπο προσέγγισης. Δεν είναι ανάγκη. Πρέπει να δούμε τη φερικιότητα δύο, αλλάζουμε τα πράγματα, ε, είμαστε με στη συζήτηση αλλά ρεαλιστικά. Δεν είναι μόνο ο τραπεζικός τομέας και θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης για το πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το, η εικόνα της αγοράς είναι πολύ πιο πιο περίπλοκη. Η ΚΕΙ έκανε μια σύγκριση, όχι, έχουμε μια αντίθεση. Είδα την αιτιολογική έκθεση και την, τα σχόλια. Υπάρχει περίπου μια κριτική της εξέλιξης της κατάστασης. Σας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούσαμε να βρούμε μια ισορροπία, αλλά να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο ε, και και ε, να μην ε, έχουμε για τις ασφάλειες αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε για τις ε, τράπεζες. Νομίζω ο Λεωνάρντο και άλλοι έκαναν σχόλια. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε προσθέτοντας μερικές τροπολογίες και σε συζήτηση μαζί σου. Αλλά ίσως να αλλάξεις και λίγο τον τίτλο σου και να έχουμε ανάκαμψη και εξυγίανση είναι τραπεζική έκφραση. Ε, ακόμα και ε, ίσως ε, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο εφόσον εδώ μιλάμε για μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι ναι. έκθεση ιδιές πρωτοβουλία, γι' αυτό μπορούμε να προσθέσουμε και ένα υπότιτλο. Κανένας άλλος δεν θέλει το λόγο. Η Κέι για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Έχω και στην προηγούμενη έκθεση, θυμάστε τον τίτλο, είχε και ένα και λοιπά στο τέλος και ούτε αυτό δεν μπορέσαμε να βγάλουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ε, για να είναι η αγορά πιο ε, στέρεα και πιο διαφανής. σε διάφορα νομοθετήματα που έχουμε ε, είτε ψηφίσει είτε είναι καθοδό έχουν πολλά ζητήματα διακυβέρνησης. Ε, και ελπίζω να ε, λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα πλέον. Δεν ξεκινούμε από μηδενική βάση, θυμίζω. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βασική δομή και υποδομή, ε, είτε ήδη στημένη, είτε καθοδόν, όπως σας είπα, προετοιμάζεται. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανάκαμψη και η εξυγίανση να καλύπτει και πιστοτικά ιδρύματα που δεν είναι τράπεζες. Όπως και αν θέλουμε να τα περιγράψουμε και να τα ορίσουμε, είναι πολύ σημαντικό σε καιρούς κρίσης να έχει συμφωνηθεί ένα θέμα κατόπιν ε, ορίμου σκέψεως για το πώς θα ε, καλύπτονται αυτές οι καταστάσεις. Να μην έχουμε ευνηδιασμούς και εκπλήξεις ε, και ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν όλα αυτά και να υπάρχει σταθερότητα γενικά στη λειτουργία των αγορών και όχι σε μεμονωμένους φορείς. Και οι αρχές ε, CPS IOSCO ε, θα πρέπει να μπουν σε αυτό το σύστημα για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Χιούμπνερ ότι χρειάζεται ε, στενή συνεργασία για την εκαθάριση μεταξύ διαφόρων κρατικών αρχών και ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός να γίνεται διασυνοριακά, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παγκοσμίω, γιατί υπάρχουν τέτοιες εταιρείε με παγκόσμια δράση. Και συμφωνώ και για με αυτό που είπε η Σάρον για το ΕΣΑ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, ε, να ε, έχει ρόλο εκεί και για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και για τους υπολείπους. Τώρα για το πεδίο εφαρμογή. ελπίζω να συμφωνήσουμε. Ε, CCP, CSD και ενδεχομένως συστήματα πλήρωμων, οι πράσινοι πρότειναν βέβαια να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή. Κοιτάξτε ποιο πρόβλημα έχω. Το είπε ο κύριος Ντομενίτσι και ο κύριος Κίνερ τώρα μόλις. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων ε, ε, μπαίνουν σε νέα επιχειρησιακά μοντέλα, είτε μας αρέσει είτε όχι, αλλάζει η αγορά, αλλάζει ο ρόλος τους. Ε, και μιλήσατε και για τη ρευστότητα και Σάρων ε, στην τιτλοποίηση και τη χρήση. Παίζουν διαφορετικό ρόλο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά και ενδεχομένως ε, χρειάζεται να μπει ξεχωριστά είτε στην έκθεση για τις ε, παρατράπεζες, είτε κάπου αλλού. Είναι τόσο μεγάλο θέμα που χρειάζεται ειδικό κείμενο, ειδική έκθεση ξεχωριστή. Και το ίδιο ισχύει για τις ασφάλειες με τη φεραγγιότητα δύο βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι μάλλον προθύστορο να αρχίσουμε τώρα να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες στη δική μου έκθεση. Γιατί η CSD και η CCP και τα συστήματα πληρωμών έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ως σύστημα και πιέζουν και πιέζονται από το ΕΜΙΡ που είναι ο κανονισμός για τις υποδομές των αγορών και άλλα νομοθετήματα Νομίζω ότι θα μπλέξουμε αν τα βερδέψουμε ε, όλα αυτά. Ε, θα προτιμούσα να έχουμε μια έκθεση πιο στοχευμένη. Δεν ξέρω, στις συνεδρίες των σχεδόν ίσως να το κοιτάξουμε αυτό για το πεδίο εφαρμογή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει... μια προτίμηση στο να εστιάσουμε περισσότερο σε κάποια σημεία παρά να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή. Ξέρω ότι είναι σημαντικά, αλλά αξίζουν ξεχωριστή έκθεση αυτά τα ζητήματα. Ε, δεν ταυτίζω τα επιστοτικά ε, ιδρύματα με τις τράπεζες, ούτε έχω πρόβλημα με όλες τις τράπεζες. Αλλά καλά είναι να τα συζητούμε και εδώ. Ορισμένοι ε, ε, πέρασαν καλά και αλόβητη σχεδόν την κρίση και θα πρέπει να διδαχθούμε και από εκείνους. Και επίσης οι φορείς χρηματαγοράς στην Ευρώπη υπάρχουν ορισμένοι που, που τα πήγαν πολύ καλά και δεν ε, εξετάζουν θέματα πτώχευσης ή συλλογικής. Τώρα μιλούμε για έκτακτες εξετάσεις, ε, καταστάσεις, ε, εξαιρετικές, θα πρέπει οι εταιρείε να σκεφτούν και τις νομικέ επιπτώσεις. Καλό είναι αυτό. Είναι απαραίτητο να τι υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο να προβλέψουν μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει η οργάνωση αυτή να διασφαλίσει τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Θα πρέπει να έχουν προβλέψει κάτι εάν συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Νομίζω ότι μετά από τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δεχτούν όλοι, δεν νομίζω να υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και όπως είπα είδα ότι ζητείτε ένα ξεχωριστό καθεστώς για τις κρίσιμες αυτές υποδομές και όχι να ενταχθούμε μόνο στα πλαίσια των πιστοτικών ιδρυμάτων. Θα γίνει μια συζήτηση ευρύτερη σε σχέση με τη διαφορά ανάμεσα στην εξυγίανση και την ανάκαμψη και σε ποιο βαθμό τίθεται επίσης και το θέμα των, των επενδύσεων των λεγόμενων πελατών στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πλαίσια πιθανώς και της δημιουργίας μιας ειδικής αρχής εποπτείας. Ε, πράγματι, αν τυχόν κληθεί ο πελάτης να συνεισφέρει, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Απαιτούνται πολλαπλή γύρια ανακεφαλαιοποίησης από τα μέλη και τα μέλη αυτά τα διαχειριστικά πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους από τους μελάτες και δεν θα πρέπει οι πελάτες να υφίστανται τις συνέπειες. Υπάρχει ένα τείχος προστασίας στο εσωτερικό του ΕΜΙΡ, το οποίο ελπίζω να γίνει σεβαστό στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών. Περιμένω τις τροπολογίες σας τον μήνα Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ λέει η κυρία Μπάουλς. Η προθεσμία είναι η 3η Σεπτεμβρίου και θα σας ενοχλήσει κατά τη διάρκεια και ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ στις 17 ε, Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα θα δώσω την Προεδρία στον Θείοντορ, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει για το υπόλοιπο πρωινό, γιατί πρέπει να προετοιμαστώ ε, για τις διοργανικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχουμε την έκθεση του Γιώργαν Κλούτε. Συγκρισιμότητα ε, στους λογαριασμούς πληρωμών. Ε, είναι το σημείο 11. Κύριε Κλούτε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι χρειάστηκε να γίνουν πολλέ απόπειρε. Ο Μισελ Μπανιέ μου είπε ότι πέντε φορέ αποπειράθηκε να το φέρει αυτό το θέμα μέχρι να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ευδοκιμήσει. Εσύ τώρα πέρασα. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω και μόνο το γεγονός ότι έφερε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά είναι πολύ καλή για την εργασία μας αλλά και για τα συμφέροντα και τα μελήματά μας και τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. 4 ε, Ιουλίου του 12 πριν από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε την έκθεση πρωτοβουλίας. Στην έκθεση αυτή πρωτοβουλίας θυμάστε πρόκειτο βασικά για τον τραπεζικό λογαριασμό ε, και την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό το είχαμε συζητήσει πολύ, ήταν και μεγάλη πλειοψηφία που το υποστήριξε στην Ολομέλεια και ελπίζω να μπορέσουμε να βασιστούμε σε αυτό και να χτίσουμε την επόμενη έκθεση. Και να βρούμε μια καλή λύση προς όφελος και των ψηφοφόρων μας και των πολιτών εν γέννη. Τι συζητούμε σήμερα, κάποιους κανόνες ε, οι οποίοι θα κρυθούν από το πόσο ενισχύουν τους καταναλωτές και τους δίνουν τη δυνατότητα ε, να ζουν σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και να τον αξιοποιούν και όλα στα τέλη για τους λογαριασμούς. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί και ε, πολλοί να επανακτηθεί η ε, εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Δεν το καταλαβαίνουμε όταν είμαστε από τη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου έχει κλονιστεί πάρα πολύ η εμπιστοσύνη στις τράπεζες υπάρχουν και χώρες που ε, ο κόσμος δεν μπορεί τα χρήματα που έχει εξοικονομήσει, αποταμιεύσει, κερδίσει, ε, να τα εμπιστευτεί σε μια τράπεζα. Διότι ακριβώς δεν εμπιστεύεται την τράπεζα για να της δώσει τα χρήματά του. Θα πρέπει λοιπόν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη γενικά ε, στο τραπεζικό σύστημα στις τράπεζες και να λειτουργεί η εσωτερική αγορά και να μπορεί ε, σε όλα τα σημεία της Ένωσης να αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς και με σωστό τρόπο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν αφορά μόνο την πρόσβαση και δεν ρυθμίζει μόνο την πρόσβαση σε λογαριασμούς, αλλά μιλάει και για τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών και για λόγους αφήνειας και ασφάλειας δικαίου όταν κάποιος αλλάζει τράπεζα. Ε, από τη μια τράπεζα στην άλλη ή αλλάζει λογαριασμό μέσα στην ίδια τράπεζα. Με τη σειρά να σας πω ποια είναι η δομή της έκθεσης. Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τα τραπεζικά τέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέσων και εργαλείων για να υποστηρίξουν τους πελάτες να καταλαβαίνουν καλύτερα τα τέλη, να μπορούν να τα συγκρίνουν και να παίρνουν αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως. Πού ανοίγουν λογαριασμό, σε ποια τράπεζα και για ποιο λόγο. Πριν ανοίξει βέβαια κανείς ένα νέο λογαριασμό, θα πρέπει οι τράπεζες να δίνουν ευρύτατη πληροφόρηση στους πελάτες για τα τέλη. Αυτό ισχύει σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες. Ε, για να ξέρει ο πελάτης ποια τέλη επιβάλλονται, σε ποιες πληρωμές ή σε ποια πακέτα λογαριασμών. Για να μπορεί να συγκρίνει ο πελάτης τις τιμές και τα τέλη θα πρέπει και η ορολογία να είναι εναρμονισμένη και για πελάτες που έχουν προβλήματα κατανόησης ε, ε, θα πρέπει να φτιάχνουν και ένα γλωσσάρι επεξηγηματικό οι τράπεζες για να μπορούν να τρέχουν οι καταναλωτές και να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Επίσης, άπαξ ετησίως ε, θα πρέπει να τους δίνεται και ένα απολογισμό των τελών που έχουν πληρώσει κατά τη διάρκεια του έτους. Για ποιο λόγο, για να μπορούν και πάλι να το συγκρίνουν με άλλες προσφορές. Και τέλος, στη χώρα του κάθε, κάθε πελάτης ε, θα πρέπει να έχει μια ιστοσελίδα που να συγκρίνει τα τέλη και να ε, είναι πιστοποιημένη, ας πούμε να υπάρχει ένα σήμα, μια σφραγίδα κάπου ότι είναι εγκεκριμένος αυτός ο ιστότοπος και ε, αξιόπιστος. Αυτό είναι το πακέτο λοιπόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι προφανή και αυτονόητα. Αν μπω σήμερα σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα, είναι φυσιολογικό να αναγράφονται οι τιμές. Α, ξέρεις, πας ένα προϊόν, πόσο κοστίζει. Γιατί να μην ισχύει αυτό και για την τράπεζα. Και να ξέρει ε, ε, τι θα πληρώνει ο καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν και οι τράπεζε προϊόντα πουλούν. Γιατί δεν είναι τα τέλη του διαφανή. Γιατί να μην ισχύει ότι ισχύει και προφανέ σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα αναγραφή τιμών επί του προϊόντο έχω και μερικές διευκρινήσεις σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις έχω στην έκθεση. Ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε λίγο τους ορισμούς. Στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών υπήρξαν κάποιες ε, διαφορές, κάποιες ασάφειες και πιστεύω ότι έχει νόημα εδώ να συμφωνήσουμε στους ίδιους ορισμούς για να καταλάβουμε ε, περί τίνος πρόκειται και να αποφευθούν παρερμηνίες και παρεξηγήσεις πριν ανοίξει λογαριασμό ένα καταναλωτή, θα πρέπει να γνωρίζει καταρχήν όλα τα τραπεζικά τέλη που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει συμπεριλαμβανομένων και ε, όλων των τόκων και των ε, εσόδων. οι ιστότοποι ε, με τις συγκρίσεις των τελών είναι χρήσιμη υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ανεξάρτητοι ε, και θα ανταποκρίνονται και σε κάποια υψηλά ε, πρότυπα ποιότητας. Και οι υποπτικές αρχές που θα πρέπει να γνωρίζουν τις εξελίξεις των τελών θα πρέπει να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και καταρχήν θα μπορούσε κανείς να αναμένει από τις επιοπτικές αρχές να προσφέρουν οι ίδιες μια ιστοσελίδα με συγκρίση των τελών, ανεξαρτήτως των ε, υπολείπων. Και πέραν της εθνικής ιστοσελίδας ε, θα πρέπει να υπάρχει και μια δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να το κάνει η ΕΜΠΑ, η Τραπεζική Αρχή, γιατί έχουμε εσωτερική αγορά, για να μπορεί ε, ο καθένας να συγκρίνει. Δεν χρειάζονται επικαλύψεις μια πύλη, να μπαίνει ο καταναλωτής και να μπορεί να έχει πρόσβαση στους ιστοτόπους ε, με ένα σύνδεσμο των διαφόρων κρατών μελών. Ένα άλλο που ενδιαφέρει την ε, οδηγία είναι πιο εύκολη αλλαγή λογαριασμού. Τι είστε αλλαγή λογαριασμού. Καμιά φορά είναι δύσκολη η διαδικασία και λεπτή. Και κάποιοι καταναλωτές διστάζουν να αλλάξουν τράπεζα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να ε, φέρει εδώ μια διευκρίνηση με προθεσμίες, γιατί πολύ συχνά αυτή είναι μια διαδικασία που τραβά σε μάκρος. Δηλαδή μια τράπεζα που χάνει ένα πελάτη ε, δεν του διευκολύνει ε, και τη ζωή και αυτό μπορεί να επιφέρει επιπλέον τέλη, επιπλέον κόστος ή αρχικό κόστος όταν αλλάζει λογαριασμό με κάποιες νέες συσκευέ στη νέα τράπεζα. Και η νέα τράπεζα θα πρέπει να αναλαμβάνει ε, την ευθύνη να ενημερώνει τον καταναλωτή και για το ΣΕΠΑ και για τα προγράμματα και τα συστήματα επικοινωνίας. Ας πούμε, εγώ ζητώ οι πελάτες που θέλουν να αλλάξουν τράπεζα και να μεταφέρουν λογαριασμό ο οποίος είναι ε, πάνω από ένα έτος στην τράπεζα αυτή να μην έχουν κανένα ε, κόστος. Βέβαια δεν θέλω να υπάρξει και τουρισμός τώρα ένα hopping από τη μια τράπεζα στην άλλη να αλλάζει ο καθένας κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες λογαριασμό αλλά αν διατηρεί ένα λογαριασμό ε, ένα έτος και μετά αλλάζει τράπεζα θα πρέπει το κόστος αυτό να το υπομίζεται η νέα τράπεζα, η οποία στο κάτω-κάτω αποκτά ένα νέο πελάτη κάτι θα πρέπει να καταβάλει και αυτή. Ε, ε, επίσης, για την ε, ενίσχυση του ανταγωνισμού ε, στις μικρές χώρες, μας ενδιαφέρει να προωθηθεί αυτό. Βλέπουμε μια συγκέντρωση τραπεζών τώρα με την κρίση, αλλά υπάρχουν και μερικά πρακτικά προβλήματα. Το συζήτησα με ορισμένους εκπροσώπους τραπεζών Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και νομικά προβλήματα ε, εκτός του χώρου ΣΕΠΑ όταν μεταφέρει κάποιος ένα λογαριασμό με ε, βάρη. Θα το συζητήσουμε αυτά εκτενέστερα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ πρακτικό και μπορούμε να βρούμε και πρακτική λύση. Αν θέλουμε λοιπόν να είναι εύκολη η αλλαγή τράπεζας, ε, μεταφορά λογαριασμού και με λιγότερα προβλήματα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά που προτείνουν ε, οι καταναλωτές. Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του τραπεζικού λογαριασμού, ε, του αριθμού του λογαριασμού, όπως είναι με το κινητό τηλέφωνο. Στη Σουηδία συμβαίνει αυτό με την ασφάλεια. Αυτό βέβαια για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις, όχι για ιδιώτες. Ε, αυτό δεν είναι βραχυπρόθεσμη, προοπτική είναι μέσο πρόθεσμη μάλλον. Να μπορεί κανείς να έχει ένα αριθμό λογαριασμού και όταν αλλάζει τράπεζα και λογαριασμό να το μεταφέρει. Ε, έχει νόημα να το σκεφτούμε, να μας απασχολήσει. Γιατί πραγματικά θα πλούστευε ε, την κατάσταση. Ή κάτι άλλο που κάνουν οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί ένα είδος μεταφοράς όλων των πληρωμών που γίνεται από ένα λογαριασμό όταν αλλάζει τράπεζα και μεταφέρεις το λογαριασμό. Δεν λέω να γίνει αύριο, αλλά και αυτό θα είχε νόημα και να, να το συζητήσουμε. Υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες, γιατί να μην τις διευκολύνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ειδικές εμπειρίες των κρατών μελών και ε, να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη, να υποχρεώσει να τα ενθαρρύνει και να τα υποστηρίξει να κάνουν αυτές τις αλλαγές σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Την πρόσβαση στο βασικό λογαριασμό το έχουμε ξανασυζητήσει στην έκθεση ιδέα πρωτοβουλία μου και συμφωνήσαμε σε ένα συμβασμό, ο οποίος είναι το κατευθυντήριο νήμα ε, και ο Ιρμός και για την ε, συγκεκριμένη μου έκθεση έχω κάνει τροπολογίες που προσανατολίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, στα όσα προτείναμε στην έκθεση πρωτοβουλίας μας. Και με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το Κοινοβούλιο οι συντονιστές συμφωνήσαμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν τις ευρωεκλογέ. Γίνεται αυτό, προλαβαίνουμε. Θέλω να το τονίσω και είναι και θέμα αξιοπιστίας μας να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε. Αυτά. Α, μια λέξη να πω μόνο για την πρόσβαση στις τράπεζες. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ε, σε σχέση με την έκθεση ε, πρωτοβουλίας εκεί είχαμε συμφωνήσει καταρχήν να ανοίξουμε όλες τις τράπεζες ή να υποχρεώσουμε όλες τις τράπεζες να διαθέτουν, να προσφέρουν ένα βασικό λογαριασμό με κάποιες ε, εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες τράπεζες όπου μπορούμε να φανταστούμε εξαιρέσεις. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε αυτό και να το επιβάλλουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγει ότι τελικά θα πρέπει μία τράπεζα να υποχρεώνεται. Δεν συμφωνώ. Ούτε διευκολύνεται έτσι η κινητικότητα και η μεταφορά των λογαριασμών δηλαδή και στο εσωτερικό της ε, ε, ενιαίας αγοράς, ούτε ε, έχει να κάνει με ίσους όρους ανταγωνισμού, αφήστε δε που κάνει και διακρίσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που για κοινωνικούς λόγους εξαρτώνται ε, από αυτή τη ρύθμιση. Δεν μπορεί να είναι μία η τράπεζα που παρέχει ένα βασικό λογαριασμό γιατί αμέσως θα φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δυσκολίες οικονομικές και κοινωνικές θα ήθελα να παρακαλέσω αυτό να διατηρηθεί που πρότεινα στην έκθεση πρωτοβουλία για όλε τι τράπεζε, με πολύ λίγε εξαιρέσει και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω και με το Συμβούλιο γι' αυτό βασικά θα συγκρουστούμε. Αυτά εισαγωγικά είχα να πω για την έκθεση. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε και με χαρά περιμένω τα σχόλιά σα και τι προτάσει. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Κλούτε πραγματικά έκανε πάρα πολλή δουλειά. και 118 τροπολογίες έχει κάνει στο σχέδιο της πρότασης. Όπως τόνισε και ο ίδιος, βασίστηκε στην πρόταση και απόφαση του Κοινοβουλίου για την πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά φαίνεται ότι ό,τι δεν είχε μπει τότε στο συμβιβασμό και είναι δική του ευθύνη, επανέρχεται σε τροπολογίε τώρα. Έχει κάνει καλή δουλειά, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους συμβιβασμούς και πώς τους στηρούμε στο διενεκές, όχι μόνο όταν ψηφίζουμε. Μετά, η διεύρυνση του θέματος. Είχαμε συμφωνήσει για πρόσβαση σε βασικέ ε, τραπεζικέ υπηρεσίε Ενδιαφέρον το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για συγκρισιμότητα τραπεζικών τελών, αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Αυτό είναι τμήμα του πακέτου για την εσωτερική αγορά, πράξη 1 και 2. Αλλά η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι από ό,τι φαίνεται τόσο απλή να εφαρμοστεί και να μεταφερθεί στην πράξη. Ε, το, αυτό το περιγράφει στη σελίδα 3 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 58 ε, εκατομμύρια πολίτες στην Ένωση δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και από αυτούς τα 25 επιθυμούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχει να κάνει πάντα αυτό με τη φερεγιότητα, με την πιστοληπτική ικανότητα ή με προσωπικά στοιχεία, αλλά έχει να κάνει και με τις παραδόσεις. Σε ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης, Ε, ο κόσμος συνδέεται πιο πολύ με τα μετρητά παρά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχει να κάνει με την παράδοση ε, και με την ε, εμπιστοσύνη και με το να διευκολύνει την πρόσβαση δεν σημαίνει ότι ανοίγουν λογαριασμό. Στη Γερμανία υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που πληρώνουν με μετρητά και το προτιμούν αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει με πώς να το πω, ότι θέλουν να αποφύγουν διάφορα πράγματα που συνδέονται με φόρους, ούτε χρήμα ξεπλένουν. Είναι παράδοση. Οι άνθρωποι θέλουν τα μετρητά. Συμπέρασμα. Η αρμοδιότητα θα πρέπει να είναι των κρατών μελών. Μόνο τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν γιατί αυτά έχουν τη δυνατότητα με συγκεκριμένα μέτρα να αλλάξουν τις συμπεριφορές και να τις βελτιώσουν. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οδηγία και συμφωνώ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο συνάδελφος Κλούτε έχει κάνει τη βασική του έκθεση και μας τη σκιαγράφησε, αλλά εγώ πιστεύω ότι σε δύο σημεία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Πρώτον, σε 7-8 σημεία της έκθεσης μιλά για επιπλέον ε, κατεξουδότηση πράξης που ζητεί ο αλλά γνωρίζουμε ότι μια σειρά συναδέλφων ε, έχουν πολύ κριτική θεώρηση η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η ΕΜΠΑ, όλα αυτά έχουν ένα γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Εγώ έχω επιφυλάξεις, πολλές και βασικές. Θα πρέπει περισσότερο να ρυθμίσουμε τα δεδομένα, τα πρακτικά, τα πραγματικά στοιχεία, οπότε δεν χρειαζόμαστε αυτές τις κατεξουδότηση πράξη. Ένα αυτό. Δεύτερο, ενημέρωση για τα τραπεζικά τέλη. Θεμητό είναι και σωστό ε, να το ζητάτε σε διάφορες τράπεζες. Αυτό ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα στη Γερμανία. Ε, υπάρχει ένας όμιλος που ε, διαφημίζει ότι οι λογαριασμοί είναι δωρεάν, τελώς, Ναι, αλλά κάπου πρέπει να κερδίσουν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει κίνδυνος ε, να μην είναι δεδομένη η συγκρισιμότητα εξού και η οδηγία. Ε, το θέμα ε, του τραπεζικού λογαριασμού που θα μπορεί κανείς να μεταφέρει. Το πρότεινε ο κύριος Κλούτε. Αλλά αυτό νομίζω ότι αντιτίθεται με το ΣΕΠΑ. Έχουμε ε, τώρα υποχρεωτικούς αριθμούς με τον εθνικό κώδικα, ένα περιφερειακό και ένα τραπεζικό, ανάλογα με τη δομή των τραπεζών στις χώρες μέλη. Και τώρα να έχουμε από τη μια τη ΣΕΠΑ με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους αριθμούς και μετά παράλληλα να στήσουμε ένα άλλο σύστημα με ένα μετοφερόμενο αριθμό φοβούμε ότι θα αυξηθεί το κόστος για το επιπλέον σύστημα. Μέχρι 15 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να φτάσει αυτό το κόστος. Με τέτοια υπερχρέωση που έχουν οι τράπεζες, ε, με τέτοιο βαθμό ε, και των μέτρων που χρειάζονται για την εξυγείαση των τραπεζών, ο κύριο Κλούτε είπε όχι αύριο, μακροπρόθεσμα, εντάξει. Αλλά έχω επιφυλάξει ε, αν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορεί να ισχύει αυτό στη Σουηδία, ενδεχομένω και με επιτυχία να γίνεται για τις επιχειρήσεις, σημαίνει ότι είναι γνώμονα για πανευρωπαϊκή εφαρμογή. Όπως και η υπηρεσία μεταφοράς ε, του λογαριασμού. Μα κατά την άποψή μου, ο καταναλωτή θα πρέπει να αποφασίζει. Τι εντολές θα δίνει σε ένα νέο λογαριασμό για να πληρώνονται από την τράπεζα αυτόματα ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί ο καταναλωτής να δίνει αυτή την εξοδότηση, ναι, αλλά όχι υποχρεωτικά, δηλαδή να παίρνουν το λογαριασμό σου όπως είναι από τη μια τράπεζα, να το μεταφέρουν με όλες τις εντολές στην άλλη τράπεζα και να πληρώνεις και από πάνω. Ε, και το τελευταίο, ή μάλλον το επόμενο, έχει κάνει πολλές προτάσεις ο κύριος Κλούτε, μεταξύ αυτών ορισμένες είναι χρήσιμες για την κοινή εξυγίαση και καθάριση, αλλά πολλές υπερβαίνουν αυτό το στόχο. Παράδειγμα, η δικτυακή πύλη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την τραπεζική αρχή, την ΕΜΠΑ. Κανονικά, ε, ο τραπεζικός λογαριασμός του κάθε καταναλωτή έχει να κάνει με τη μητρική του γλώσσα. και μόνο το 0,27 των καταναλωτών έχουν ε, ε, διεθνή λογαριασμό ή λογαριασμό σε άλλη χώρα. Εγώ έχω λογαριασμό στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στη Γερμανία, εντάξει, αλλά είμαι προβουλευτής ε, και θέλω να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες επιτόπου. Αλλά αξίζει τον κόπο όλη αυτή η φασαρία με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή που προτείνει ο κύριος Κλούτε είναι όφελος αυτό για τον καταναλωτή ή μήπως υπερβολή που θα οδηγήσει σε υπερβολικό κόστος χωρίς πραγματικό όφελος. Γιατί με προβληματίζει αυτό. Ε, το θέμα της εξουσίας ε, ρύθμισης και η Επιτροπή το λέγει και ε, υποστηρίζει και επιβεβαιώνει και τον κύριο Μπαρνιέ ότι οι πρώτες απόπειρες όλες απερίφθησαν από την ε, Επιτροπή για τη Μελέτη Αντικτύπου, δύο μάλιστα, αρχικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνέχεια κάναν και άλλες αλλαγές και ξανάφεραν την πρόταση και ακριβώς για αυτή τη συνολική επίπτωση υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνούμε όλοι με την απόφαση του Ιουλίου του 2012 ότι ε, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό με διαφάνεια, με συγκρισιμότητα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μέτρα ε, που τα δικαιολογεί η εσωτερική αγορά χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και παρακαλώ τον κύριο Κλούτε, ε, τον οποίο σέβομαι και τιμώ για το ζήλο του, 2 Σεπτεμβρίου προθεσμία νομίζω είναι εχθρική προς τις ελληνές διακοπές. Ε, έχουμε πολλή δουλειά στις διακοπές. Τώρα επιβαρύνουμε και τους βοηθούς και τους ε, ενεργάτες. Μην βάζετε τόσο φιλόδεξη προθεσμία. Το Κοινοβούλιο έχει ολομέλειες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και τα λοιπά μέχρι τον Απρίλιο. Το, πολύ, το νωρίτερο 15 Σεπτεμβρίου παρακαλώ, όχι 2 Σεπτεμβρίου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. δείχνεται επικοδομητικό πνεύμα επί της ουσίας και εμείς άλλωστε θέλουμε μια σωστή οδηγία και λογική, αλλά να μην οδηγήσει και στην πλήρη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Λούντβικσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εν πάση περιπτώσει, τον εισήγητη και πράγματι πολλά από τα θέματα τα οποία θέτει είναι πολύ σημαντικά. Επί τη βάση της έκθεσης πρωτοβουλία που είχαμε υιοθετήσει το 12, συνεχίζουμε να εργαζόμεθα. Υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία το 12 γύρω από το θέμα αυτό και έτσι μπορούμε με την ίδια λογική να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Η συζήτηση μέχρι τώρα μετά την πρόταση της Επιτροπής ζητά ε, την, ε, επικαλείται μάλλον την αρχή της επικουρικότητας. Έχω όμως την αίσθηση ότι στο παρόν πλαίσιο η ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία εν πολλής είναι αρκετά τεκμηριωμένη. Ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ο καθένας για την επικουρικότητα. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια καταναλωτών στην Ευρώπη, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να έχουν στη διάθεσή τους ένα τροπόζικο λογαριασμό, τον οποίο δεν μπορούν να έχουν. Αποκλείονται από την αγορά λόγω ε, υψηλών κειμενωμένων τελών και επίσης πάρα πολύ ε, ακριβό είναι το να αλλάξει ε, κανείς λογαριασμό. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό το να αλλάξει τράπεζα και λογαριασμό. Και οι δυσκολίες αυτές ε, απαγορεύουν ουσιαστικά τη σωστή ανάπτυξη της ενίας αγοράς και την κινητικότητα. Άλλωστε και το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα καθυστερεί στην ανάπτυξή του και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει υψηλότερη διαφάνεια και ενημέρωση για το κόστος της αλλαγής λογαριασμών και της αλλαγής τραπεζών. Μέχρι τώρα το πρόβλημα αυτό της αλλαγής λογαριασμού ή του ανοίγματο λογαριασμού δεν έχει αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει συνεπώς να μας απασχολήσει το θέμα και πολλά είναι αυτά τα οποία μένει να βελτιωθούν ακόμα. Δεν είναι λογικό ε, στην παρούσα φάση να ισχύει η κατάσταση που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο. Θα συνεισφέρουμε λοιπόν στην ε, επεξεργασία της έκθεσης αυτής με μεγάλη ταχύτητα έτσι ώστε να γίνει συνολικά δεκτό. Πρέπει να υπάρχει αναγνώριση του δικαιώματος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει το σύστημα αυτό να ισχύει για όλους τους ε, που έχουν την δυνατότητα αυτή και θα πρέπει οι τράπεζες να υπακούν σε βασικούς κανόνες στα πλαίσια του συστήματος πληρωμών. Ένας βασικός λογαριασμός, η έλλειψη ενός τέτοιου βασικού λογαριασμού μπορεί να στιγματίσει επίσης αυτούς οι οποίοι δεν τον έχουν και είναι ιδιαίτερα λυπηρό οι λιγότερο ελκυστικοί καταναλωτές να αποκλείονται από υπηρεσίες όπως οι συγκεκριμένες πιστοτικές υπηρεσίες. Το θέμα δεν είναι να διευρύνουμε μια κατηγορία πελατών που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις έτσι ώστε οι τρέχοντες λογαριασμοί να φέρουν εις πέρα συγκεκριμένε αποστολές και σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς να παρέχονται κάποιες βασικές υπηρεσίες. Και έτσι θα μειώσουμε και το κόστος. Θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι τα ε, τέλη για τους βασικούς ε, απλούς λογαριασμούς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει απλότητα και να είναι εύκολη κατανοητή η λειτουργία των λογαριασμών και να μην περιπλέκονται τα πράγματα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά περίπλοκη. Μην ξεχνάμε ότι οι ρυθμίσεις τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχουν στο στόχο την απλούστευση της ζωής των καταναλωτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το τέλος, τα τέλη και να έχουν τις ε, τραπεζικές υπηρεσίε. Το να απαιτούνται μεγάλοι κατάλογοι εγγράφων, τεκμηρίων κτλ. είναι κάτι το οποίο δεν ε, θα συνεισφέρει στην δημιουργία της απαιτούμενης διαφάνειας. Απαιτείται λοιπόν οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες οι οποίες συνοδεύουν έναν απλό ε, τραπεζικό λογαριασμό να είναι απλές και κατανοητές. Σχετικά τώρα με την αλλαγή, την δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού, εδώ θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με δύο διαφορετικούς τρόπους σχετικά με τους χρονικούς λογαριασμούς, δηλαδή κάθε πότε θα μπορεί κάποιος να αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό από τη μία τράπεζα στην άλλη. Και από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει ένα διακανονιστικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη έτσι ώστε σε εθνικό επίπεδο να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις στην περίπτωση αλλαγής λογαριασμού. Η δυνατότητα αλλαγής θα πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει να μπορεί να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για την αλλαγή λογαριασμών οι οποίοι σήμερα ισχύουν και εφόσον θεωρούνται θετικοί μπορεί να αποτελέσουν τμήμα του συστήματος στο μέλλον. Απαιτείται πάντως μεγάλη διαφάνεια και γνώση των συνθήκων αλλαγής απαιτείται γνώση του συνολικού κόστους και απαιτείται επίσης και γνώση σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κάτι το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον είναι οι διαμεθοριακές αλλαγές. Ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται στην αλλαγή των τραπεζών μια χώρα η οποία δεν ανήκει στο ευρώ, είναι εκτός της ζώνης ευρώ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια βήματα προς τα εμπρός Πρέπει να διασφαλίσουμε την κινητικότητα και πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτά είναι τα προκαταρκτικά σχόλια τα οποία έχω να κάνω. Πάντως μας έχει δώσει μια πλήρη πρόταση, σωστά επεξεργασμένη και από κοινού θα προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε και να καταλήξουμε στις σωστές συμβιβαστικές λύσεις που θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας. Thank Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φιλίπ Ντεμπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κλούτε ε, για όλη την εργασία που κατέβαλε και στο παρελθόν επίσης όταν ήταν μεταξύ αυτών που εργάστηκαν για, ήδη για έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό και βασίζουμε την εργασία μας πάνω στα όσα είχαν γίνει προηγουμένως σε αυτήν την Επιτροπή και στην έκθεση που είχε δημοσιευτεί. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι μια καλή πρόταση διότι ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που υπάρχει. Το μόνο που θα ήθελα να κάνω στην αρχή αυτής της συζήτησης είχα αναφέρει ε, την, ε, την διάκριση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αφενός ε, μιλούμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό, όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά συστήματα πληρωμών για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα εσωτερικής αγοράς συνόρων. Οι ανάγκες που έχουν αυτοί δύο αυτές ομάδες ατόμων είναι διαφορετικές. Στην αρχή λοιπόν τη συζήτηση θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε και τα δύο προβλήματα, τα προβλήματα των δύο αυτών κατηγοριών και πρέπει να κάνουμε διάκριση. Επίσης, στόχος μας πρέπει να είναι διτός από την άποψη αυτή. Συζητούμε επίση τα βασικά συστήματα πληρωμών, προσπαθώντα να, να μην έχουμε κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, προσπαθώντα επίση να επιλύσουμε προβλήματα εσωτερική αγορά και τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν πολλοί που είναι εδώ, οι όσοι εργάστηκαν στο παρελθόν ή θα εργαστούν στο μέλλον πάνω σε αυτό το θέμα, έχουμε τον ίδιο στόχο. Η μόνη συζήτηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς θα επιτύχουμε το στόχο που επιδιώκουμε όλοι. Υπάρχουν μερικές ιδέες που έχω σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής και την πρόταση του κυρίου Κλούτε. Πρώτα απ' όλα σχετικά Καμιά φορά ξέρουμε ότι ε, ε, μέσα στα κράτη-μέλη για να αλλάξουμε τράπεζα ε, χρειάζεται χρονικό περιθώριο και κόστος και πρέπει να δούμε ότι αυτή η μεταφορά να μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα κυρίως μεταξύ των κρατών μελών διότι συνήθως τώρα η μεταφορά γίνεται μεταξύ κρατών μελών και θα πρέπει να προχωρήσουμε βασιζόμενοι στην προγενέστερη έκθεση. Επίσης η διαφάνεια των τελών είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ξέρουμε εξάντε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις συναφείς υπηρεσίες το κόστος για ε, τον καταναλωτή. Συζητήσαμε στο παρελθόν, Βεβαίω δεν πρέπει να είναι δωρεάν οι υπηρεσίες, θα πρέπει να έχουν μια τιμή, αλλά δεν μπορεί να είναι υψηλότερο το, η τιμή από ό,τι σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν συστήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη, ε, ε, ε, οι διάφορες οργανώσεις, αφιλοκερδείς οργανώσεις για πληρωμές σε διάφορες χώρες. Θα πρέπει να καλύψουμε τις, μη, αυτές τις, μη, τις, τις οργανώσεις, αυτές τις φιλανθρωπικές ε, οι οποίες θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ξέρουν πολύ καλά τι πληρώνουν, να υπάρχει διαφάνεια. Ο κύριος Κλούτε επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση του συστήματος και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, στην αρχή του πακέτου, να υπάρχει ε, σαφής ένα σύνολο υπηρεσιών σε μια, με ένα δεδομένο κόστος. Έτσι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το θέμα της τυποποίησης είναι επίσης έχει βαρύνουσα σημασία. Δεν είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέα ορολογία, αλλά θα πρέπει να εναρμονίσουμε ορισμένα όρους που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη για να υπάρχει εκεί ε, σαφήνεια και διαφάνεια, γιατί αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουμε. Ο κύριος Κλούτε πρότεινε επίσης ε, τα βασικά ε, να μεταφέρεται ε, ο αριθμός του εμβάσματος και αυτό είναι κάτι δύσκολο να γίνει, δεν ξέρω αν αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης αναφέρθηκε ο κύριος Λάγκες, αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε εδώ ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν θα είναι, που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι μεγαλύτερα από τα προβλήματα που θα επιλύσουμε. Γενικά νομίζω ότι η εισήγηση εδώ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Βεβαίως θα έχουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, συνηγορό υπέρ του γεγονότος να έχουμε μια φιλόδοξη εισήγηση που να περιλαμβάνει ε, την, ε, την συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς ε, κοινωνικούς και οικονομικούς και επίσης να καλύπτεται αυτό διασυνοριακά διότι πάρα πολλοί νέοι φοιτητέ και άλλοι που αναζητούν εργασία ε, διασχίζουν τα σύνορα και θα πρέπει να καλυφθούν από ε, τραπεζικής πλευράς ω προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς και οι υπηρεσίες να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια και θα πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν φιλοδοξία στο θέμα αυτό και ελπίζω να έχουμε έτσι μια πολύ καλή εισήγηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολτ τώρα. Έχω πολλά να προσθέσω. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ε, χαιρετίζω το γεγονός ότι η εισήγηση αυτή έχει υποβλήθει. Ε, περιμέναμε πολύ καιρό αυτή την εισήγηση. Ανέφερε, επισήμανε τα προβλήματα ο εισήγητής που συνήντησε και ο Μίσελ Μπαγνιέ επίσης στην Επιτροπή είχε προβλήματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ε, προσθέσουμε, να μην ενισχύσουμε ε, το συνέστημα ότι η Ευρώπη ε, ενδιαφέρεται μόνο για τις επιστοληπτικές οργανώσεις, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές όταν πρόκειται για τα προβλήματα των πιο αδύναμων που δεν μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό ή να κλείσουν ένα λογαριασμό που είναι δαπανηρός, ότι δεν ενδιαφερόμαστε εμείς. Σχετικά με το θέμα αυτό, εμείς, όπως είπε ο Φίλιπ Ντεμπάκερ, έχουμε μια φιλόδοξη εισήγηση και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι οι λύσεις στις διάφορες χώρες ίσως φαίνονται διαφορετικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ουσιαστική προσέγγιση και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για ένα πράγμα. Αυτό είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις αυτή η προσφορά τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί για να, να μην χρησιμοποιείται για να γίνεται διάκριση ε, και ε, να μην δίνει ένα σήμα στον καταναλωτή που είναι ορατός στους τρίτους. Αυτό θα αποδυνάμωμε τους αδύναμους αντί να τους ενισχύσει. Θα ήταν ηρωνικό εάν το γεγονός ότι μερικοί πρωταγωνιστές. Μερικοί εμπλεκόμενοι εργάζονται με τους φτωχούς όπως μερικές οργανώσεις πιστωτών, μερικά ταμιευτήρια στις χώρες μας. Το γεγονός ότι ήδη προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιείται ως λόγος, ως αιτία του ότι άλλοι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Βεβαίως το πνεύμα αυτών των ενώσεων, των πιστοτικών, το αρχικό δεν ήταν να πούν ότι τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Οργανώθηκαν επειδή οι τράπεζες δεν συναλλασσόντουσαν με όλους, με όλους όσοι, όσους θα έπρεπε να συναλλάσσονται. Θα πρέπει λοιπόν να ενδιαφερθούμε για τους πιο αδύναμους, τους πτωχούς ε, πελάτες, όχι μόνο εμείς αλλά και όλες οι τράπεζες. Δεν ζημιώνουμε την Deutsche Bank ανασχοληθεί με κάποιον που έχει ένα χαμηλό βασικό εισόδημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και από την άποψη του ανταγωνισμού. Τέλος, υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο δεν άκουσα ακόμη μια καλή λύση. Δηλαδή, εάν διευκολύνουμε για καλούς λόγους την μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών, διότι αυτή θα είναι η καλύτερη μέθοδος και η ολιγότερο παρεμβατική να μειώσουμε το υπερβολικό κόστος των τραπεζικών λογαριασμών. Αν το θέλουμε αυτό, το πρόβλημα είναι ότι αν οι συγκριτικοί πίνακες, ιστότοπους κλπ. συγκρίνουν μόνο το κόστος, εμείς βεβαίως θα μπορούσαμε να παροτρύνουμε τις τράπεζες να υιοθετήσουν ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα, να συγκρίνουν την Apple με χλάδια, να συγκρίνουν το μήλο με το χλάδι. Ε, αν έχουν ένα μεγάλο δίκτυο υποκαταστημάτων, ενώ άλλες απλώς εργάζονται διαδικτυακά. Αν συγκρίνουμε τα δύο, ε, όταν έχετε μια ανοιχτή γραμμή και όταν έχετε ένα άτομο με το οποίο μπορείτε να συζητήσετε και παρέχει υπηρεσία στην κοινότητα, τότε μπορείτε να συγκρίνετε χλάδια με μήλα. Και τότε ε, τα συγκριτικά μέτρα πρέπει να προσέξετε ούτως ώστε να μην επιφέρουν διακρίσεις εναντίον αυτών που παρέχουν επίσης ένα ε, σύστημα δικτύων υποκαταστημάτων ή άλλες ε, βελτιώσεις ε, ποιοτικέ. Υπάρχει βεβαίως και το πρόβλημα του τι γίνεται με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Να απλώς συγκρίνεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανεξάρτητα του εάν η τράπεζα έχει μεγάλο ή μικρό κεφάλαιο. Αυτό οθεί μερικά επιχειρηματικά μοντέλα όπου μπορούμε να έχουμε λιγότερου κεφαλαϊκούς πόρους, ενώ άλλες τράπεζες την χάνουν καλύτερης διαχείρισης και εμφανίζονται ως να είναι ίδια τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα. Αν δούμε ε, ότι έχουμε ένα μπεϊλίν 100.000 ε, ε, ευρώ, αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή. Τα εγγυημένες αυτές οι καταθέσεις, ακόμα και αν έχουν περισσότερα χρήματα, παρόλο που αυτοί είναι λίγοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εάν ε, περάσουμε σε αυτό την προσέγγιση της σύγκρισης, το κριτήριο για τη σύγκριση δεν θα πρέπει, να είναι μόνο το κόστος αλλά και η ποιότητα. Και εκτός αυτού είναι σημαντική ιδέα ούτως ώστε να αυξήσουμε τη, διασυνοριακή δραστηριότητα, να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει αυτό με κριτήρια αμφισβητήσιμα. Νομίζω εκτός αυτών ότι η εργασία του Κλούτε είναι πολύ καλή, έχει καλό προσανατολισμό, αλλά θα πρέπει εδώ να εργαστούμε το συντομότερο δυνατόν, διότι ο στόχος θα πρέπει να είναι στον κατάλογο των νομοθετημάτων που θα περάσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον κάτι που να στοχεύει ε, στους αδύναμους στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Με συγχωρώ να πω ότι έχουμε ήδη έναν κατάλογο συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο και ζητώ από όλους σας που θα λάβετε το λόγο να προσπαθήσετε να είστε πάρα πολύ σύντομοι, διότι έχουμε ήδη περιορισμένο χρόνο. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κάμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο αυτό που εκπώνησε τόσο γρήγορα. Σημερίζουμε ορισμένες ανησυχίες των άλλων σκιωδών και του εισηγητή. Νομίζω ότι ο Φιλίπ έχει δίκιο όταν λέει ότι ότι μιλάμε για πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πολλοί δεν έχουν πρόσβαση. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα διαφωνούσε κανείς με την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση. Ε, ε, ε, το θέμα της ε, νέας αγοράς επίσης, τα θέματα σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διάφορα επίπεδα, ε, διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δεκτοί οι πελάτες. Ο πατέρας μου ήταν από μια κοινότητα μεταναστών και αυτή η κοινότητα αποκλειόταν, δεν ήταν κοινότητα που γινόταν δεκτή στις τράπεζες και στις πιστοτικές κάρτες. Ε, ε, ε, ζούσε μόνο με ρευστά και δεν είχε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, διότι με την τεχνολογία ίσως κανείς δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό, αλλά μπορεί να έχει πιστοτική κάρτα. Ακόμα και αν έχει τραπεζικό λογαριασμό, μπορεί να, έχει, να αγοράζει στο ίντερνετ, να αγοράζει προϊόντα, διότι έχουμε αυτά τα μέσα τα τεχνολογικά. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε ότι ας μην έχουμε αυτήν την συζήτηση μιλώντας πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερες κασέτες και δίσκους και CDs στην εποχή του MP3 και του MP4. Οι τράπεζες δεν έχουν ε, εξαλείψει τα παλιά μοντέλα Βεβαίως, έχουμε την ηλεκτρονική τραπεζική, έχουμε την τραπεζική διατηλεφώνου, αλλά ε, οι τράπεζες τι κάνουν, ε, ε, ε, έχουν, έχουν τους πιστωτές, τους οι οποίοι διασταυρώνονται και μια εναλλακτική θα ήταν τεχνολογικά να σπάσει αυτό το μοντέλο. Ξέρω ο Σβέν μίλησε για σύγκριση μεταξύ μήλων και αχλαδιών, αλλά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το μήλο το Apple. Αλλά πρέπει να εξετάσετε τι θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία σε μας. Κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ανησυχώ πάρα πολύ ότι προσπαθούμε να αναγκάσουμε τις τράπεζες να, και προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τραπεζών στην αγορά όταν έχουμε ε, διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Ε, θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για τράπεζες που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες με τις πιστοτικές οργανώσεις διότι θα καταλήξουμε με μια κατάσταση όπου αυτοί που θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες θα έχουν την χειρότερη υπηρεσία διότι τους σωθήσαμε σε αυτήν την αγορά και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφουμε τις πιστοτικές οργανώσεις καλύπτοντας ένα κενό στην αγορά. Θα πρέπει αυτοί οι εναλλακτικοί πιστωτές να τους καθοδηγήσουμε και βλέπω στη δική μου την εκλογική περιφέρεια δεν πρέπει ε, να δώσουμε τόση πολλή εξουσία στις τράπεζες ώστε άλλοι άλλοι να αποκλειστούν. Μετά έχουμε το θέμα της ενίας αγοράς. Θέλουν οι άνθρωποι όντως να μεταφέρουν τους λογαριασμούς από μια χώρα στην άλλη. Αυτό εξαρτάται βεβαίω από ποια χώρα προέρχεστε. Πολλοί νέοι στη χώρα μου λένε ότι αυτό που θέλουμε είναι όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό για ένα έτος να μπορούμε να ανοίξουμε ένα λογαριασμό εκεί ε, και να μεταφέρουμε χρήματα και όχι να περνάμε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Γαλλία, στη Γερμανία και μετά να επιστρέφουμε. Έχουμε εδώ ένα πραγματικό πρόβλημα. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερή είναι αυτό και μετά έχουμε τη διαφάνεια ένα από τα μεγάλα θέματα διαφάνειας και δύο είναι τα σημαντικά στις τράπεζες είναι ε, τα ε, απατηλά, ε, απατηλές ανακοινώσεις σχετικά με τα επιτόκια. Μερικοί βλέπουν έναν αριθμό και δεν καταλαβαίνω. Ένας φίλος μου άφησε 100 λίρες στο ένα φίλο του και του είπε θα με, πληρώσετε σε, με πληρώσεις σε δύο, σε δύο εβδομάδες 110 δάνεισε στο φίλο του δάνεισε 100 λίρες σε κάποιον που έπρεπε να το επιστρέψει σε λίγο χρονικό διάστημα 110. Ε, αλλά βεβαίως αυτό ε, είναι αν θέλετε ένα στοκογλύφος, αλλά αν δείτε τους αριθμούς τους ίδιους 100 λίρες και επιστροφή 110 μετά από δύο εβδομάδες, ε, τι γίνεται με την διαφάνεια πόσο πρέπει ε, αυτό με τις τράπεζες, τι γίνεται με μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο. Ε, νομίζω ότι αυτό επιτρέπει την σύγκριση αν έχουμε κάποια διαφάνεια. Δύο και το τελευταίο πράγμα για την διαφάνεια. Έχουμε διαφάνεια ε, σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα τραπεζικών λογαριασμών. Όταν κανείς καταθέτει λεφτά σε μια τράπεζα, δεν μένουν τα λεφτά στην τράπεζα. Πιστώνει, ε, δανείζει σε μια τράπεζα ο καταθέτης, ο οποίος ε, δανείζει τα χρήματα αυτά και παίρνει μεγαλύτερο υποτέκιο. Θα πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν είναι η τράπεζα που κρατάει την κατάθεση, αλλά δανείζει τα χρήματα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάμπο. Ο κύριος Μπάλτς και παρακαλώ όλοι να τηρείτε το χρόνο σας, να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι, έχουμε χρονικό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τον εισηγητή μας τον Γιώργιον Κλούτε ο οποίος πραγματικά επέδειξε πολύ μεγάλο ζήλο και επιμέλεια και ε, ασχολήθηκε με όλα τα θέματα και τα έχει συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αντιλέγει αυτή, σε αυτή την πρόταση. Ο κόσμος μάλλον χαίρεται που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και κάνουμε και την πρόταση και παίρνουμε την πρωτοβουλία. Πλην όμως έχει σημασία να δημιουργήσουμε και τις σωστές προϋποθέσεις να σταθμίσουμε με προσοχή τα υπέρ και τα κατά πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα. Και όπως ε, με όλα μας τα νομοθετήματα να έχουμε και το σωστό μέτρο πάντα υπόψη μας. Ε, σύντομες παρατηρήσεις για τα πεδία εφαρμογής. Η ρύθμιση για την πρόσβαση ε, στο λογαριασμό πληρωμών για όλους είναι κάτι που βλέπω έτσι με κάποια επιφύλαξη στο μέλλον οι καταναλωτές ανεξαρτήτως ε, χώρας προέλευσης και ε, τόπου κατοικίας να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν λογαριασμό όπου επιθυμούν. Όχι στη χώρα τους, όχι στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό με βρίσκει κάπως διστακτικό. Πώς θα μεταφραστεί και θα εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά σε ποιο βαθμό μπορεί να ελεγχθεί ο καταναλωτής πριν να ανοίξει το λογαριασμό. Γιατί δεν υπάρχουν ελάχιστε απαιτήσει όπως είναι το εισόδημα ή ε, η κατοικία. Ο βασικός λογαριασμός επίσης ε, δεν θα πρέπει να έχει δυνατότητα να περνάει στο κόκκινο, δηλαδή να έχει αρνητικό υπόλοιπο. Δεν είναι ένας μηχανισμός δανεισμού. Και να πω κάτι επίσης και για την αναλογικότητα, ε, όπως σε όλα τα νομοθετήματα μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές αυτό το θέμα. Ξέρω ότι ε, δεν πρόκειται όλες οι τράπεζες να θυγούν από ένα τέτοιο βασικό λογαριασμό. Είναι μάλλον οι τοπικές τράπεζες, οι εγχώριες και ε, ε, έχει εύκολη πρόσβαση ο καθημερινός άνθρωπος. Αυτό όμω μπορεί να σημαίνει και μεγαλύτερη γραφειοκρατία και διοικητικό άχθος για τις τράπεζες αυτές. Και ακριβώς όταν είναι μικρή η τράπεζα δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα. Σε άλλους τομείς και πεδία εφαρμογή υπάρχουν ε, καλές προτάσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ε, Κλούτε, περισσότερη διαφάνεια για τα τραπεζικά τέλη, αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ήδη μεγάλη διαφάνεια, για να μην πω μέγιστη, σε αυτά τα θέματα και δεν θα πρέπει να χαθούν αυτά τα καλά που ισχύουν. Αυτό ισχύει επίσης και για την αλλαγή λογαριασμού. Αν μπορεί ο καθένας να ανοίγει ένα βασικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης, ε, θα προϋποθέτει και μεγάλη κινητικότητα των καταναλωτών αυτό. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν είναι εύκολη, απλή αλλαγή λογαριασμού από μία τράπεζα σε τράπεζα σε άλλη χώρα. Το κόστος θα πρέπει να είναι αρκετά έτσι, σε ένα πλαίσιο και ε, το διοικητικό βάρος για τις τράπεζες. Επίσης για την πρακτική εφαρμογή πρέπει να ρυθμιστούν ακόμα ορισμένε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Οι επόμενοι συνάδελφοι μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Ιντβελτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ο οποίος δημιούργησε μια εξαιρετική βάση για τη συζήτηση που ακολούθησε. Είναι χαριτωμένος ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε μέσα, τα οποία ισχύουν εδώ και αιώνες θα έλεγα, και όπως είπε ο προηγούμενος συνάδελφος ο κόσμος παρόλα αυτά αναπτύσσεται με τρομερές ταχύτητες και τα μέσα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα ξεπερασμένα. Και γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κ. Ντεμπάκερ, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και όχι να εμένουμε στις παραδόσεις. Θα πρέπει να δεχτούμε τις αλλαγές γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει εν δεν κουβαλάμε σακούλες ε, ε, με νομίσματα και δεν κουβαλάνε τα μουλάρια τα επιταγές πάνω από τα βουνά πλέον αλλά παρόλα αυτά οι αγορές εξακολουθούν να είναι ε, πιστεύουν ορισμένοι εθνικές και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, θέλουμε να αναπτύξουμε και την διαδικασία την αντίστοιχη με τις Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό καθιστά επίγον το να έχουμε μια πραγματική ενιαία αγορά, όχι τις οικονομίες 28 μελών που να συνεργάζονται. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν τις, τους πιστοτικούς λογαριασμούς και ε, διαμεθοριακά και να κρατούν τον αριθμό τον οποίο πάντα είχαν. Αυτό μπορεί να γίνεται και γίνεται σε εθνικό επίπεδο και ελπίζω και σε διεθνές επίπεδο. Στα κινητά τηλέφωνα αλλάζει εταιρεία αλλά κρατάς τον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο είχες. Ένα αντίστοιχο σύστημα θα μπορέσει να υπάρξει και για τις τράπεζες. Είμαι βέβαιος ότι με ε, τα, ένα απλό σύστημα ανταλλασσομένων με περιπτώσει νομισμάτων θα μπορέσουμε να βρούμε μια κάποια λύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εφόσον θέλουμε να αναπτύξουμε μια εσωτερική αγορά και για, το λιανικό, ε, για τις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των νέων συστημάτων και δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, δεσμευτικοί ε, και αρνητικοί. Πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι λοιπόν και να κάνουμε ένα θετικό βήμα έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε λογαριασμούς, να μπορούμε να αλλάζουμε διαμεθοριακά λογαριασμούς και να κρατάμε και τον παλαιό αριθμό. Ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτής της συζήτησης υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το ένα υπάρχει το, της συμπερίληψης στο πιστοτικό σύστημα και εδώ θα συμφωνήσουμε με τις περισσότερες προτάσεις που έκανε ο εξαιρετικός εισηγητής μας. Και από την άλλη υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ο εξυγχρονισμός του πιστοτικού κόσμου. Να μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες είναι μια βιομηχανική δραστηριότητα και δεν βρισκόμαστε σε ένα σύστημα κατευθυνόμενης οικονομίας. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε την ελεύθερη αγορά από τη μία και από την άλλη να επιβάλλουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν κόστος στους εμπλεκομένους, στον παραγωγό ιδιαίτερα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί γιατί επιβαρύνοντας τις πιστοτικές εταιρείες σε επενδύσεις και σε κόστη έτσι ώστε να περάσουν σε νέες τεχνολογικές καταστάσεις αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες όπως κανόνες ασφαλείας, περιβαλλοντικοί κανόνες και έχω την εντύπωση ότι το θέμα της διαμεθοριακής αλλαγής λογαριασμών δεν είναι κάτι το άμεσα προβλέψιμο. Θα πρέπει να το κρατήσουμε για το μέλλον, αλλά πιστεύοντας ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα. Ε, και όσο επίσης πιέζουμε προς την online πιστοτική δραστηριότητα τόσο λιγότερες θέσεις απασχόλησης θα έχουμε στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά την οποία έχει επιτελέσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ ε, συμμερίζομαι αυτά που είπε ο Λάγκια να μην χαλάσουμε τις διακοπές μας, αλλά πρέπει να δώσουμε μια γρήγορη απάντηση γιατί το κείμενο είναι σημαντικό. Ό,τι έχουμε κάνει για τις αγορές, για το ΕΜΙΡ είναι όλα καλά, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο λοιπόν να διαφωνούμε, αλλά εδώ και κάποιες δεκαετίες προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αν επιβάλλουμε κάποια λογικά πράγματα στις τράπεζες, όχι υπερβολικά, σαν παράδειγμα τη συγκρισιμότητα των τελών. Δεν θα πάθουν και τίποτα σοβαρό και νομίζω ότι ο πιστωτικός τομέας είναι αυτός για τον οποίο οι πολίτες δεν θα κλάψουν ιδιαίτερα αν τυχόν τους επιβάλλουμε κάτι. Λοιπόν, ε, διαφάνεια είναι απαραίτητη, ε, το είπαν πολλοί αυτοί, για να γίνονται σωστές επιλογές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι. Είναι αλήθεια ότι προς στιγμή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους διαμεθοριακούς λογαριασμούς, αλλά αναπτύσσεται το να ζει κανείς σε πολλές χώρες. Ότι όλα αυτά ήταν σπάνια πριν 20 χρόνια, ενώ είναι πολύ συνηθισμένα τώρα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για αυτούς που έχουν προβλήματα. και να διευκολύνουμε επίσης ε, τις ε, διαμεθοριακές τραπεζικές εργασίες. Ε, νομίζω ότι έτσι θα αποφύγουμε επίσης και το να στιγματίσουμε ε, τις, ε, τους πολίτες οι οποίοι έχουν προβλήματα σε σχέση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι ότι οι πολίτες θέλουν να έχουν κάποιες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες σε καταστάσεις ισότητας και όσο ασχολούμαστε περισσότερο με τους καταναλωτές χωρίς να κάνουμε διακρίσεις τόσο το καλύτερο. Μια αντιμετώπιση λοιπόν που θα επιτρέψει σε όλους να βρουν κάποιες λύσεις με πλαισιωμένες ε, φυσικά προσφορές υπηρεσιών διότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες και πρέπει να είμαστε και αρκετά φιλόδοξοι γιατί η πολυδιάσπαση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην κρίση δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Υπάρχει το θέμα των ψηφιακών πληρωμών σαν παράδειγμα που θέλουμε να προωθήσουμε και ευχαριστώ ε, τον Γιούργεν και να του πω ότι του έχουμε κάθε εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Επιστρέφω τώρα στον κύριο Κλούτε. Παρακαλώ να είστε σύντομο. Ο κύριο Λάγκεν. Μια παρατήρηση να κάνω μόνο για τη Σοφή Γκουλάρ. Όχι, τη, τη Σοφή Νετβέλτ, συγγνώμη. Ε, Σοφή είναι η Νετβέλτ. Εμένα με λένε Σιλβί, λέει η κυρία Γκουλάρ. Ναι, εντάξει, στην κυρία Νετβέλ απευθύνομαι. Ε, ζήτησε ε, μια εσωτερική αγορά πλήρη. Αυτό δεν εξαρτάται τώρα από το βασικό λογαριασμό αν θα ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να διατηρηθεί η αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη για το βασικό λογαριασμό. Ε, η μεταφορά, η ΣΕΠΑ, τα τέλη, εντάξει αυτά είναι σημαντικά και σημαντικότερα για την εσωτερική αγορά παρά η ε, απόλυτη ελευθερία και δυνατότητα να έχει κανείς ένα βασικό λογαριασμό όπου επιθυμεί, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, εισοδήματος, κύκλου γνωριμιών, φίλων κτλ. Ωραία. Ε, ο συγητής έχει το λόγο. Παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε σύντομος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, τους συναδέλφους για τα όσα είπαν. Νομίζω σε γενικές γραμμές συμφωνούμε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σας είπα ότι είμαι πρόθυμος και για ρεαλιστική πρόσβαση. Αυτό το τελευταίο, το ένα σημείο του Βέρνερ Λάγκερ πρέπει να το συζητήσουμε εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τις λεπτομέρειες ίσως χρειαστεί να τις συζητήσουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά το να αφήσουμε απολύτω αυτό το θέμα στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών με βρίσκει και μένα επιφυλακτικό, γιατί δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζες ότι αναγνωρίζεται ένα λογαριασμό ανεξαρτήτως χώρα. Διότι άκουσα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ζεις και σπουδάζεις είσαι υποχρεωμένος να έχεις στη Μεγάλη Βρετανία λογαριασμό και δεν αναγνωρίζουν το γερμανικό σου λογαριασμό. Αν αναγνωρίζουν το γερμανικό σου λογαριασμό λύνεται το πρόβλημα. Ναι, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη λύση. Κουνάει το κεφάλι του κ. Λαν. Αυτά. Όταν έρθουν οι τροπολογίε θα έχουμε την ευκαιρία να τις συζητήσουμε και να περάσουμε και συμβασμούς. Ένα σημαντικό ρώτησε ο κύριος Λάγκεν, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα. Επίτηδες το βάλαμε τόσο σφιχτό. Ακριβώς απλούστατα για να έχουμε μια δυνατότητα να το ολοκληρώσουμε πριν τα τέλη του έτους και, ή της θητείας, εν Από την άλλη, βέβαια, το ξέρω ότι επηρεάζει τις διακοπές. Να αλλάξουμε κατά μία εβδομάδα να, να παρατείνουμε. Δεν ξέρω, πρόεδρε, τι λέτε. Ε, αναβολή, παράταση της προθεσμίας ε, κατά μία εβδομάδα. Σχετικά με την πρόταση χρονοδιαγράμματος, θα εξετάσουμε το αίτημά σας για την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης και αυτό θα επηρεάσει το σύνολο του χρονοδιαγράμματος. Θα σας επιβεβαιώσουμε όμως το τι μπορεί να γίνει μέσω ε, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πάντως να είσαστε πάρα πολύ σύντομος γιατί έχουμε και άλλη μια έκθεση παρακαλώ. Εγώ τελείωσα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και παίρνουμε στην τελευταία έκθεση για ε, το πρωινό. Είναι της κυρίας Φερέιρα. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών Εφαρμογή των Προτεραιοτήτων για το 2013. Δίνω μέσα στο λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά για πιο γρήγορα. The 2013 semester cycle. Uh, and it represents the European Parliament's input on lessons to be learned uh, for the next semester. Σχετικά με τα μαθήματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε για το επόμενο εξάμεινο. Είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα επί τη βάση των συστάσεων για τις συγκεκριμένες χώρες, των συγκεκριμένων αναχώρα συστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί συνάδελφοι διάβασαν την έκθεση και εγώ θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στις βασικές ιδέες σας. Νομίζω ότι οι συστάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά δεν έχει υπάρξει πάρα πολύ σημαντική κίνηση. υπάρχουν κάποια απλά μηνύματα τα οποία μπορούμε, στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε πέρα από την δημοσιονομική εξυγίανση που είναι φυσικά βασικό. Έχουμε αρκετή εμπειρία λέξη πλέον για να κατανοήσουμε ότι αν δεν υπάρξει μια ελάχιστη ανάπτυξη δεν θα, να, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη εξυγίανση των δημοσιονομικών. Ξέρετε τι έγινε στην Πορτογαλία με την παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών όπου ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι συστάσεις της Τρόικα. Στην επιστολή την οποία απέστειλε ο τέος Υπουργός Οικονομικών δείχνει ότι στην Πορτογαλική περίπτωση τα μέτρα λιτότητας τα οποία εφαρμόστηκαν δεν του επέτρεπε να πετύχει τους στόχους τους οποίους είχε και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο κατέθεσε την παρέτησή του. Ένας από τους λόγους, ίσως ο πιο σημαντικός. Απαιτείται πραγματική ανάπτυξη, λοιπόν είναι απαραίτητη η ανάπτυξη για να αποκατασταθεί η ισορροπία των δημοσίων λογαριασμών και του ε, προϋπολογισμού της κάθε χώρας. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα έτσι ώστε συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα να τεθούν σε πρακτική το ταχύτερο δυνατόν. Όλοι το λένε, στα λόγια όλοι αυτό πετυχαίνουν υποτίθεται, αλλά στην ουσία τίποτα. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν για την αποτυχία αυτή, ποιες είναι οι αιτίες, ποιες είναι οι αιτίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε αυτήν την ανάπτυξη και πώς μπορούν ε, ίσως ε, οι, ε, οι χώρες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τη ζήτηση μέσω αύξησης ε, σταδιακά ε, τους μισθούς και έτσι να αναπτυχθεί η οικονομία και να τραβήξει και τις υπέλπες χώρες ε, με έναν συμμετρικό τρόπο όπως ακριβώς κάνουμε και με τις χώρες οι οποίες είναι ελληματικές οι οποίες στην ουσία περιορίζουν την εσωτερική τους ζήτηση. Δεν μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε την αντιμετώπιση του ενιαίου μοντέλου για όλους. Υπάρχουν διαφορετικές συστάσεις γιατί οι διαφορετικές εθνικές οικονομίες θα πρέπει να προσαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο και κάτω από διαφορετικά οικονομικά πρότυπα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως να ενισχύσουμε την αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ. Γιατί οι χώρες οι οποίες ανήκουν σε ένα ενιαίο χωρονομίσματος δεν έχουν τα παραδοσιακά μέσα του μηχανισμού των συναλλαγμάτων και των εθνικών ανεξάρτητων λογαριασμών για να δώσουν κίνητρα στην οικονομία τους. Δεν έχουν τους μηχανισμούς αυτούς. Είναι απαραίτητο λοιπόν ότι αν επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας ηφεσιακά ε, σε όλες τις χώρες τότε ε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχουν οι συγκεκριμένες οικονομίες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλες τις πληροφορίες που έχουμε και στο μηχανισμό προειδοποίησης, έγκαιρης προειδοποίησης. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναλύσει με ε, αναλυτικό τρόπο τις ασυμμετρικές επιπτώσεις που υπάρχουν στις διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες μετά από την εφαρμογή των ομοιογενών πολιτικών στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ζητάμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια προσεκτική αξιολόγηση των προσδοκιών ανάπτυξης, έτσι όπως παρουσιάζονται, έχουν αρκετή εμπειρία σε σχέση με τις προβλέψεις τους, τις οποίες αναθεωρούν προς τα κάτω βέβαια, και αυτό δημιουργεί άγχος στους πολίτες και ιδιαίτερα στους επενδυτές. Πρέπει λοιπόν να, να ελέγξουν την ποιότητα των προβλέψεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε ε, αυτά τα οποία κάνουμε ε, να μην λειτουργούν αρνητικά. Θα πρέπει επίσης ε, να επενδύσουμε στην παραγωγικότητα, στην εκπαίδευση και στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και να μην ξεχνάμε και την Ευρώπη για 2020. Οι στόχοι 2020 για την Ευρώπη του 2020 δεν έχουν προχωρήσει αποτελεσματικά εφόσον θέλουμε εμείς ε, να λειτουργήσουμε σαν ε, μελλοντικός αποτελεσματικός εταίρος. Χρειάζεται να επενδύσουμε λοιπόν σε τομείς οι οποίοι να διασφαλίσουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Και ζητάμε παράλληλα κάποιες πρωτοβουλίες ε, να συντονιστούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έτσι ώστε να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση. Πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα στήριξη των κρατών μελών που καλούνται να εφαρμόσουν τις διαφορετικές αλλαγές τις οποίες τους έχουμε συστήσει. Περιμένουμε λοιπόν για μια πρωτοβουλία η οποία έχει επανειλημμένα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το μέσο CCI ανταγωνιστικότητα και σύγκληση. Και περιμένουμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, να αξιολογήσει το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής, όπως επίσης και σε επίπεδο εξωτερικής εμπορικής πολιτικής που να μην βασίζεται στον προστατευτισμό αλλά σε αυξημένες ανάγκες αμοιβαιότητας για να διευκολύνουμε τις προσβάσεις σε τρίτες αγορές που είναι και αυτό απαραίτητο για να αναπτυχθούμε. Ζητάμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και κάποιες εκ των προτέρων αξιολογήσεις των κοινωνικών επιπτώσεων όλων των προτινομένων μεταρρυθμίσεων και διαφορετικών αλλαγών και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και μέσω του κοινωνικού πυλώνα μετά από αυτά στα οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα πλαίσια της εκθέσεως της και η χρήση άμεσων θα έλεγα σταθεροποιητικών μέσων μερικές φορές μπλοκάρονται στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα στα οποία υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και μέσω των διαδικασιών μακροπρόθεσμων ανισορροπιών. Εν πάση περιπτώσει έχω έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας ε, η οποία είχε συμφωνηθεί μετά από τη συμφωνία για το διπλό πακέτο για το Τούπακ. Στόχος είναι να αναλυθούν οι τρόποι μέσω από τους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε μια δυνατότητα κοινή διαχείρισης του δημοσίου χρέους. Γιατί τώρα είναι σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, τα οποία βραχυπρόθεσμα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό εμείς με ευρωπαϊκό τρόπο, με σφαιρικό τρόπο. Γιατί μα μην ξεχνάμε ότι το χρέος αυτό είναι φυσικά σε ευρώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο καλεί την ολοκλήρωση τάχιστα της τραπεζικής αγοράς και της ενιαίας εποπτικής αρχής. Περιμένουμε και τη δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ταμείου, θα δούμε τι θα βγει και επίσης το σύστημα εγγύησεως των καταθέσεων. Τώρα έχουμε κάποιες βελτιώσεις στα πλαίσια του καθορισμού του τρόπου λειτουργίας και δημιουργίας ε, του συγκεκριμένου αυτού συστήματος εγγυήσεων ε, και να βοηθήσουμε επίσης ε, να ανακάμψει η οικονομία μέσω και της τελευταίας οδηγίας και να νοικοδομήσουμε την εσωτερική αγορά. Καλούμε επίσης για βήματα δράσης εναντίον της φοροαποφυγής επί τη βάση και των προηγούμενων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητάμε παράλληλα να υπάρξουν βελτιώσεις ε, του υπολόγου και του τρόπου λειτουργίας ε, της Τρόικα και την εμπλοκή του Κοινοβουλίου και σε άλλους τομείς ε, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης και την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και τα οποία δυστυχώς έχουν αρχίσει να περνούν σε διακυβερνητικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάτι το καινοτόμο σε όλα αυτά τα μηνύματα στα οποία αποστέλουμε, αλλά υπάρχει μια σειρά θεμάτων ε, για τα οποία επιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα οποία δεν έχει ακόμα πετύχει κάτι. Είναι λοιπόν χρήσιμο να προωθήσουμε τα θέματα αυτά και να ε, μετατραπούν όλα αυτά τα θέματα από λόγια σε έργα γιατί από μόνα τους δεν θα φτιάξουν τα πράγματα. Προσπαθώντας λοιπόν να έχουμε μια ευρύτερη πρόταση στη διάθεσή μας, μπορούμε να σχολιάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως να βοηθήσουμε τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Σκιώδης. Ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Φερέρα που ετοίμασε αυτήν την καλή έκθεση σχετικά με το εξάμεινο. Εμείς επαναλαμβάνουμε, όχι εκείνη, εμείς επαναλαμβάνουμε εδώ και μήνες και εξάμεινα και χρόνια τις ίδιες λέξεις. Ζητούμε την ανάπτυξη, το τέλος της λιτότητας, την αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών, κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Δεν πράττουμε τίποτα για να γίνει αυτό. Διότι νομίζουμε ότι μιλώντας απλώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά μιλώντας δεν επιλύουμε τα πρόβλημα. Ε, ψευδόμαστε στους πολίτες, στους Ευρωπαίους λέγοντας ότι τελείωσε η κρίση, ότι όλα θα βελτιωθούν. Είναι λάθος αυτό το βλέπουμε για χώρες που κατέβαλαν προσπάθειες. Η Πορτογαλία βλέπουμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χτες ρώτησα τον κύριο Ντράγκη για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει στην Πορτογαλία και είχα την τύχη να μην λάβω ε, καμία απάντηση. Και όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μέλος της Τρόικας. Θα πρέπει να είναι λίγο υπεύθυνη σχετικά με τα όσα συμβαίνουν όταν πρόκειται για νομοθετήματα, ξέρουμε ε, να τα εκπονούμε, να τα μπλοκάρουμε στο Συμβούλιο και να μιλάμε για το 2020, αλλά είμαστε ήδη στο 2013, ε, σύντομα το 2014, στα μισά του δρόμου. Πού βλέπουμε ε, τα, τους στόχους 2020 να πραγματοποιούνται. Όταν ορισμένες χώρες μιλούν για οικονομική διακυβέρνηση, οι ίδιοι αμφισβητούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό μετά επικύρωση από το Συμβούλιο. Υπάρχει θέμα συνεκτικότητας. Μας λένε συνεχώς ότι χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο καθένας αφήνει τους άλλους να πιστεύουν ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές και εξηγεί στους πολίτες, όπως γίνεται στην Γαλλία, ότι θα μεταρρυθμίσουν τις συντάξεις, αλλά δεν θα, ή δεν θα κάνουν κακό, αλλά κάνουν κακό, είναι επιζήμιες όπως μια οικογένεια που ζει κάτω από τα δυνατότητές της, πρέπει να πάρουμε μέτρα για να βρούμε κάποια σταθερότητα και για το σκοπό αυτό πρέπει να προσέξουμε τις δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες, να είναι αποτελεσματικές, να μεριμνήσουμε γι' αυτό και σε αυτούς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη που όλοι θέλουμε, δηλαδή τις επιχειρήσεις, να τους δώσουμε το πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν με εμπιστοσύνη. Μας λένε συνεχώς ότι πρέπει να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη. Πώς να αποκατασταθεί με συστήματα που αλλάζουν κάθε έξι μήνες, όπου, τα οποία συνεχώς αλλάζουμε και τροποποιούμε. Όταν κανείς αρχίζει μια επιχείρηση θέλει να ξέρει ε, πώς, ποια θα είναι η αντιμετώπιση ε, στις επόμενους μήνες, στους επόμενους πέντε μήνες. Και αυτό που λείπει σήμερα δεν είναι οι ιδέες, είναι η δραστηριότητα. Διότι την ανάπτυξη θα την ξαναβρούμε μόνο αν υπάρχει δραστηριότητα, ε, μέσα έμμεσα-μέσα. Βεβαίω λένε ότι αυτοί που είναι οι πλουσιότεροι πρέπει να ξοδεύουν περισσότερα. Σπάρουμε τη Γαλλία που γνωρίζω καλύτερα. Όταν στην αρχή τη σχολική χρονιά δίνει κανεί ένα πριμ στι οικογένειε, ε, τότε διαπιστένουμε αμέσως στα μεγάλα μαγαζιά μια αύξηση των ε, πωλήσεων των τηλεοράσεων. Πού κατασκευάζονται οι τηλεοράσεις εκτός Ευρώπης. Πρέπει να προσέχουμε τα χρήματα που κατασκευαζονται οι τηλεοράσει εκτό Ευρώπη πρεπει να προσεχουμε τα χρηματα που δινουμε ε, για την ανάπτυξη που ξοδεύονται θα έπρεπε να έχουμε μια ανάπτυξη εξθετική και αυτό δεν λειτουργεί με όλα αυτά που κάνουμε. Και αυτό σήμερα που πρέπει να περιμένουμε από αυτούς που είναι δίθεν ηγέτες είναι να δώσουν λύσεις θαραλέες. Εγώ συμβάλλω όσο μπορώ μιλώντας για την νομική ασφάλεια, ε, την φορολογική ασφάλεια, την κοινωνική ασφάλεια. Έθεσα μια δεύτερη ερώτηση στον κύριο Ντράγκη, το ρώτησα πώς υπόψη την αθλειότητα, την κοινωνική στους συστημικούς κινδύνους. Και εδώ δεν έλαβα απάντηση. Είτε είναι κανείς αριστερά είτε δεξιά, δεν μπορεί να, να μην είμαστε ευαίσθητοι σε αυτούς που βρίσκονται σε ένδια, που δεν έχουν πια τίποτα. Ασχολούμεθα με τους Αμερικανούς και ε, τι άλλο υπάρχει σε αυτό το εξάμεινο ελπίζω ότι θα έχει μερικά θετικά πλεονεκτήματα. Εκτιμώ το ότι η Κομισιό έκανε συστάσεις πιο ακριβείς, το είχαμε ζητήσει. Και Ταυτόχρονα οι συστάσεις ε, βεβαίως όταν γίνονται πιο ακριβείς λέμε ότι η Κομισιόν προχωράει πάρα πολύ αλλά δεν είναι η Κομισιόν, είναι το Συμβούλιο που πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν, αν ξαναβρούμε πραγματική δραστηριότητα και όχι τεχνάσματα οικονομολόγων που περνούν το χρόνο τους ε, λέγοντας ότι λυπούνται για τις κακές προβλέψεις τους, για δείτε το ΤΑΦ τι συμβαίνει όταν ένα μέλος της Τρόικα λέει «κάναμε λάθος», Είχαμε κάνει υπολογισμού που ήταν εσφαλμένοι. Τι θα πρέπει να πει ο ασθενή αν ο χειρουργό του είπε ότι έχω ε, ε, κάνει την ίδια εγχείρηση 10 φορέ, πέτυχα 8 φορέ, ελπίζω ότι για σένα θα είναι ή θα έχει καλό αποτέλεσμα και όχι κακό. Εάν λοιπόν ο προβληματισμό για το εξάμεινο μπορεί να καταλήξει σε κάτι το πιο συγκεκριμένο, θα πρέπει να είμαστε ευτυχεί, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν θα είναι η περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες δεν βλέπω κανένα. Ε, καλά, η κυρία Φερέιρα είναι, ναι, συγγνώμη. Ε, λέει στη συγγήτρια. Φιλελεύθερη, ουδής, ε, θέλει να μιλήσει, Οι παρόντες έχουμε. Ωραία, θα δώσω το λόγο τότε στον κύριο Λάμπερτς. Δεν το ζήτησα. Α, κοιτάξτε για αλλαγή να μιλάσω γαλλικά. Ζαμπόλ για σένα το κάνω. Συμφωνώ αρκετά μαζί σου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ανακτήσουμε ένα νέο οικονομικό στόχο και μια δυναμική στην Ευρώπη με συγκεκριμένες προτάσεις. Ελπίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου λέγοντας ότι αν στην κοινωνία στραγγαλίζουμε τους πιο αδύναμους, για να το πω απλά, δεν είναι καλύτερο. Ε, και στραγγαλίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις και τους πιο αδύναμους καταναλωτές. Ναι, το ξέρω, δεν είπα εγώ αυτό, λέει ο κ. Γκοζέ. Εντάξει, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε μια νέα δυναμική και ανάκαμψη στην οικονομία, χρειάζεται σε βάθο φορολογική μεταρρύθμιση, με κοινή δράση όμως, ευρωπαϊκή. Γιατί και πάλι αν μείνουμε σε μια φορολογική κούρσα μεταξύ μα, την πληρώνουν οι μικρή και οι μεγάλοι τη γλιτώνουν και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις εταιρείε χρειάζεται μια ελάχιστη εναρμόνιση αν όχι ολοκλήρωση σε προλογικό επίπεδο. Παρένθεση ήταν αυτή, γιατί αυτό σκέφτηκα ακούγοντάς. Ε, θα μπορούσαμε να δράσουμε εκεί, το προτιμώ συμφωνώ με την εισηγήτρια σε κάποια σημεία να τονίσω μόνο τι θέλουμε εμείς να ενισχύσουμε. Για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τι παρατηρούμε, γιατί είναι και καινούργια άσκηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάμεινο το εξάμεινο βελτιώνεται η δουλειά που γίνεται. Ε, δηλαδή, στην αρχή, από το πρώτο εξάμεινο που ήταν αμυγός κάτι της ε, Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υπόθεση. Σιγά σιγά έχουμε περάσει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ξέρουμε όμως και ότι μεταξύ διαφόρων αδελφών μερικά αδέλφια είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα και όλες οι γενικές διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ίσες. Κυριαρχεί και πάλι εκφύν σε σχέση με την απασχόληση ας ε, Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξή. Υπάρχουν ε, ειδικέ ομάδες αναχώρα και εργάζονται ε, με διαφορετικές προδιαγραφές. Να πάρω ένα παράδειγμα στην τύχη. Ας πούμε, έρευνα και ανάπτυξη. Τι δαπανούν εκεί οι χώρες. Έχουμε ένα στόχο για τη στρατηγική 2020, 3%. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό και θα μπορούσε ε, αυτό να κάνει την οικονομία μα ξανά ανταγωνιστική, αλλά τι βλέπουμε. Ορισμένες συστάσεις αναχώρα το λαμβάνουν πολύ περισσότερο αυτό υπόψη, ενώ κάποιες άλλες πολύ λιγότερο. Και περιέργως δεν έχουν τις πιο σκληρές συστάσεις οι πιο ε, κακοί μαθητές. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είμαστε σωστοί στην ε, προσέγγισή μας. Ε, θα πρέπει να συντονίσουμε τη μεθοδολογία μας ανατομία και αναχώρα για να ενισχυθεί η διαδικασία. Οπότε η νομοθετική πρόταση που εξαγγέλλεται για την εξάντε ε, συντονιστική προσπάθεια της οικονομικής πολιτικής είναι καλό, με στάνταρ και πρότυπα μεθοδολογικά κοινά. Λοιπόν, επευκαιρία, δεν ξέρω αν παρευρίσκεται κάποιος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, ελπίζω τουλάχιστον να τα διαβιβάσετε αυτά στο φίλο μας όλοι ρε, ότι το περιμένουμε και για δύο σημεία να δούμε τι θα κάνει. Πρώτον, είχε εξαγγείλει μια άσκηση για τον έλεγχο της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών. Έτσι το βαφτίζουν αυτό συχνά. Δηλαδή πώς μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα ε, τις δαπάνες, τι εστί επενδύσεις ε, μακροπρόθεμες και τι εστί λειτουργικές δαπάνες που μπορούν να εξορθολογιστούν. Μας έχει στείλει σχετική επιστολή ο κύριος Όλι Ρεν, αλλά ε, παρά είναι ισχνή. Ένα άλλο που περιμένουμε να μας απαντήσει είναι η ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θυμίζω ότι στα πλαίσια του εξαπλού πακέτου του Six Pack, στις μακροοικονομικές ισορροπίες, οι ανισορροπίες τονίσαμε ότι ενδεχομένως κοινωνικές παράμετροι μπορούν να αποτελούν σοβαρές ανισορροπίες και οικονομικές και να διακυβεύουν την οικονομική υγεία ε, των κρατών μελών και της ΟΝΕ. Άρα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό στο, ε, στη φαρέτρα μας ας πούμε να έχουμε και κοινωνικούς ε, δείκτες για να κατανοούμε τι συμβαίνει στη χώρα. Θέλουμε να δώσουμε μια νέα δυναμική, δεν είναι με 25, 26, 27%, 28 φτωχών στην Ευρώπη. Δυστυχώ αυτό συμβαίνει όμω, Κάθε χρόνο προστίθεται μία ποσοστιαία μονάδα του πληθυσμού κάτω από το όριο τη στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και πάλι μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι είναι ηθικό αυτό και ιδεολογικό πρόβλημα, γιατί εγώ είμαι από εκείνου που παίρνουμε σοβαρά την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων ότι όλοι γεννιόμαστε ίσοι και ε, ε, δεν μπορούμε το 1 τέταρτο του πληθυσμού να είναι τόσο εξαθλειωμένο ότι 100% ε, της ενέργειάς τους την αφιερώνουν στην επιβίωση. Ξεχάστε τα ηθικά και τα διοντολογικά. Είναι και ε, ανόητο εξουδετερώνεις ένα ανθρώπινο δυναμικό που ε, μόνος του αντικειμενικό σκοπός είναι να καταφέρει να επιβιώσει. Πάει χαμένη αυτή η ενέργεια. Ένα άλλο σημαντικό αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αθεκτικότητα στην οικονομία μας, θα πρέπει να δούμε και την παραγωγικότητα της εργασίας. Ανέκαθεν το λέγαμε αυτό, δεν το αμφισβητούμε, βέβαια να δούμε την παραγωγικότητα του κεφαλαίου και των πόρων. Δηλαδή, αν δούμε ε, την ε, απόδοση του κεφαλαίου και τις τιμές που πληρώνουμε για την ενέργεια και για τους φυσικούς πόρους, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολλά για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και πώς να το πω, να ε, εξημερώσουμε τους μετόχους που πρέπει να μάθουν να ζουν σε έναν κόσμο που έχουν μειωθεί τα έσοδα. Έχει δίκιο ο Ζανπόλ Γκοζές. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να μάθουν να ζουν σε έναν κόσμο που δεν πέφτουν τα λεφτά από τον ουρανό, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το ίδιο όμως ισχύει και συχνά είναι οι ίδιοι για τους μετόχους. Απόδοση 8, 10, 15, 20 το χρόνο δεν υπάρχει σε μια οικονομία της αγοράς και θα πρέπει να μάθουν να ή να ξαναμάθουν να ζουν με αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο κοινωνική δικαιοσύνη, είναι οικονομική αποδοτικότητα. Η Κίνα σχεδόν δεν επιβραβεύει το κεφάλαιο, δεν έχει καμία απόδοση. Καλά, αυτοί το παρακάνουν κιόλας. Αλλά εμείς έχουμε κέρδη από το κεφάλαιο πολύ ψηλότερα από ότι ε, αποδόσεις που είναι αξιοπρεπείς και ρεαλιστικές σε μια ε, ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε χρήματα και πόρους για τις επενδύσεις, δεν θα πρέπει να ε, επιβραβεύουμε τους ραντιέριδες, γιατί αυτό το εισόδημα δεν συνάδει με την οικονομία της αγοράς. Γι' αυτό που έλεγε η περί δημοκρατικού ελέγχου, για την ε, Τρόικα και εγώ παρακολουθώ αυτούς που λέγουν ναι, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση και ε, οικονομική στην Ευρώπη και όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι κάνουν πίσω. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε και ε, την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτου. Για να μπορέσει ο μέσος πολίτης στη Γαλλία, στο Βέλιο και αλλού να δεχθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, θα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να έχουν μια ποιότητα δημοκρατικής νομιμότητας εξίσου υψηλή είτε προέρχονται από τις Βρυξέλλες είτε από το Παρίσι. Δηλαδή εγώ πώς απαντώ σε αυτό το γεγονός ότι σήμερα δουλεύουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο που δεν έχει απαραίτητη ε, δημοκρατική νομιμότητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το καταργήσουμε. Όχι, χρειάζεται και οικονομική και πολιτική ολοκληρωσία αλλά να έχει την ίδια δημοκρατική νομιμοποίηση με εκείνη των κρατών μελών. Τούτου λεχθένους δεν είναι από εκείνους που λέγουν ότι ό,τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη ε, είναι απολύτως ε, δημοκρατικά σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Όχι. Και στο Παρίσι Ατελής είναι η δημοκρατία, όπως και στις Βρυξέλλες. Άρα, να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνεται. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος Έπινγκ. Και σας παρακαλώ να τηρήσετε το πεντάλεπτο στην τοποθέτησή σας. Ε, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω ε, σε διάρκεια αυτά που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος και θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο αργά για να διευκολύνω τη διευμηνία. Κυρία Φερέιρα, δεν έχουμε συμφωνήσει σε πάρα πολλά πράγματα και το ίδιο ισχύει και για τη συγκεκριμένη έκθεσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το πάθος το οποίο επιδείξατε βέβαια, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία διαφωνούμε και τα οποία θα προσπαθήσω να αλλάξω. Να σταθώ λοιπόν σε κάποια πιο συγκεκριμένα. Ζητάτε να υπάρξει επίγουσα εφαρμογή του CCI επί τη βάση της κοινοτικής μεθόδου. Μιλάμε για τις δημοσιονομικές δυνατότητες που θα οδηγήσουν ε, σε μια νέα μορφή οικονομία στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αντί να μάθουμε δηλαδή από τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει μέσω αυτής της οικονομίας μεταφοράς, Τώρα προσπαθούμε να επαναλάβουμε τα λάθη αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εισηγήτρια επίσης στα συμπεράσματά της ζητά να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και για τον φόρο των οικονομικών χρηματοδοτικών υπηρεσιών ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εμείς ήμασταν και σαν πολιτική ομάδα κατά του FTT ε, γιατί είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στον ανταγωνισμό. Και στο τέλος ε, μιλά τη συμπλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με ένα κοινωνικό πυλώνα και μέσω ενός πίνακα αποτελεσμάτων. Και διαρωτάτε ποιος είναι ποιο είναι το κατάλληλο όργανο για να ασχοληθεί με αυτή την πολιτική. Και είπε επίσης ότι οι πλεονασματικές χώρες θα πρέπει να προωθήσουν την εσωτερική ζήτηση για να βοηθήσουν τις άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι χώρες όπως ε, η Γερμανία τιμωρούνται γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικές. Η έκθεση λοιπόν της κυρίας Φερέιρα ε, στην ουσία είναι ανάποδη από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά στον κύριο Γκίγκολτ. Ναι, θα ήθελα να κάνω μερικές σύντομες ε, παρατηρήσεις στα γερμανικά. Εμείς οι πράσινοι τώρα μιλούμε γερμανικά κυρίως για τον Ζων Πολ Γκοζές. Σε σχέση με αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι είναι δύο πράγματα που πρέπει να διαφεροποιήσουμε. Υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες σχετικά με την οικονομική πολιτική. Ποιες είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Ορισμένοι θα πούν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυστηρή γραμμή, ανταγωνισμός ε, φορολογικός, ανταγωνισμός στους ρυθμίσεις, οικονομία της αγοράς με διαφορές σημαντικές ε, στους ε, συντηρητικούς και στους φιλελεύθερους υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις και στους σοσιαλιστές ε, θέλουμε επίσης την ανάπτυξη. Και θέλουμε την προσέγγιση των οικονομικών πολιτικών. Εξαρτάται περί τίνος πρόκειται. Ιδαλλιώς είμαστε πολύ κοντά με τους σοσιαλιστές. Βεβαίως μπορούμε πάντοτε να αγωνιζόμαστε για την ισία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ υπάρχει ένα συμβιβασμό ε, της Επιτροπής, η Στρατηγική Ευρώ 2020 ε, και η πολιτική, ε, η κοινωνική. Αλλά η Κομισιόν είναι τυφλή κάπου κάπου εδώ. Οι συνεργάτες μας στο Κοινοβούλιο λένε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για το στόχο των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας και η Εστονία εδώ έλαβε συστάσεις ενώ άλλες χώρες που ε, αδιαφορούν για την ενέργεια ε, δεν κάνουν τίποτα στις συστάσεις. Το είπε και ο Φιλίπ, στην καταπολέμηση της φτώχειας είναι πολύ λιγότερες οι συστάσεις σε σχέση με την απασχόληση. Είναι μονομερές αυτό και ασυνάρτητο γιατί δεν δίνουν συστάσεις χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά ανάλογα με το γραφείο κάθε χώρας και τις προσφυλής του Ασχολίες και τα θέματα έχουν συντάξει τις συστάσεις. Δεν είναι πετυχημένη η συνοχή του κειμένου. Υπάρχει αυτή η μονομέρεια επί της ουσίας, αλλά και το άλλο είναι ένα μεθοδολογικό ζήτημα. Και τι εννοώ. Κανείς θα πρέπει να περιμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κριτήρια τα ίδια για όλες τις χώρες για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής αν ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί να κάνει ένα απολογισμό και τις συστάσεις που απορρέουν και όχι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε desk ας πούμε της κάθε υπηρεσίας για κάθε χώρα ε, και τι αρέσει περισσότερο. Ε, ε, αυτή τη συνοχή δεν την έχουμε και τη ζήτησε πάντα ανέκαθεν το Κοινοβούλιο δεν διαφωνούμε μεταξύ μας και αυτό που με εξοργίζει ακόμα περισσότερο είναι κάτι άλλο έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα, εφαρμόζονται. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί επί τη ουσία με μεμονωμένε συστάσει, θα πρέπει να απαιτεί ε, κανεί ε, με διαφάνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ενημερώνει για το ποιε συστάσει εφαρμόζονται και ποιε όχι. Πάνω από 140 συστάσει, μόνο σε 17 έχουν γίνει μεγάλε πρόοδοι, πλήρη εφαρμογή. Αυτό το μέτρησαν οι συνεργάτε μα. Είχαν την υπομονή να το κάνουν. Ούτε καν 15% δηλαδή. Το υπόλοιπο. Ε, παρουσιάζεται με διάφορες αποχρώσεις, ε, με διάφορες ε, διευκρινήσεις στην έκθεση αναχώρα. Με καμία σαφήνεια όμως, ποια χώρα με μετέφερε ποια, με πίνακα δηλαδή. Πόσε συστάσει πήρε κάθε χώρα, ποιε εφήρμοσε, με ποιο τρόπο. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τολμά να ανταποκρίνεται στο καθήκον τη να έχει διαφάνεια για το ποιο εφαρμόζει αυτά που έχει αποφασίσει το ίδιο το Συμβούλιο. Δεν το καταλαβαίνω. Εμεί έχουμε προειδοποιήσει, έχουμε κάνει φασαρία και προσωπικά το έχω ξανασυζητήσει με ε, προσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βοηθάει αυτό τίποτα φοβά, φοβούνται να φέρουν το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών του. Το ίδιο το Συμβούλιο τα έχει αποφασίσει αυτά. Ανεξαρτήτως τώρα κομμάτων και προτιμήσεων, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής είναι τόσο σημαντικός, είναι υποχρεωμένος να πετύχει. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε χρόνο. Δώστε παρακαλώ το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί δεν τα εφαρμόζει όλα αυτά. Παρόλο που τα λέει και στι συστάσεις του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα τελευταία εξάμεινα. Και μάλιστα έχουμε προειδοποιήσει. Θέλω να μας δώσουν εδώ δημόσια στην Επιτροπή μας. Okay. Um, it seems that there is... Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο μέλος του Κοινοβουλίου που να ζητάει το λόγο. Από την Επιτροπή ίσως. Okay. Πολύ καλά. Σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ευχαριστώ, σχετικά με το θέμα της εφαρμογής φεσταμένων ε, ε, ε, συστάσεων ειδικών για τις χώρες θα ήθελα να επισύρω την προσοχή του αξιοτήμου μέλους για την, στην αξιολόγηση της Κομισιόν βεβαίως συμμεριζόμαστε το θέμα ότι δεν υπάρχει επαρκής εφαρμογή σε ορισμένους τομείς. Σε ορισμένους τομείς υπήρξε εντυπωσιακή πρόοδος ενώ σε άλλους όπως ε, είπε και ο κύριος Γκίγκολντ, έχουμε απογοητευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μια εκτίμηση της εφαρμογής μόνον ε, με βάση συγκρίσεως του αριθμού ε, υψηλής εφαρμογής κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών, όπου ο συνολικός αριθμός συστάσεων είναι την να υποτιμά ορισμένες από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Μπορούμε να πούμε ότι ενώ μοιραζόμαστε, συμμεριζόμαστε τις βασικές ανησυχίες, σημειώνουμε ότι όλα τα ε, κράτη-μέλη σε όλους τους τομείς έχουν κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ε, παροτρινόμενοι από τις συμβουλές και τις συστάσεις των θεσμικών οργάνων. Ακόμα και αν κρίνουμε ότι είναι ανεπαρκείς οι προσπάθειες, θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις του εξαμήνου υπήρξαν ε, θετικές ε, με βάση ε, τις συστάσεις για πλήρη εφαρμογή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ναι, ναι. Ο κύριος Κίγκολτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να σας πω πολύ ομά ότι δεν με ικανοποίησε η απάντησή σας. Εγώ ήμουν πολύ συγκεκριμένος στις ερωτήσεις. Αν κοιτάξετε τις διάφορες εκθέσεις αναχώρα που έχετε δημοσιεύσει, σε ορισμένες εκθέσεις μιλάτε για ευρεία εφαρμογή. Σε άλλες λέτε ε, σημαντική πρόοδος, αλλού έχει γίνει κάποια πρόοδος. Εάν συγκρίνετε την ορολογία, και το έχω κάνει εγώ και το έχουμε κάνει για όλες τις χώρες, χρησιμοποιείτε διαφορετική διατύπωση για να περιγράψετε αν οι χώρες έχουν κάνει πρόοδο, μεγάλη, μικρή, λίγο, πολύ κτλ. Ε, ε, ουσιαστικά τι κάνετε. Είναι αδύνατο να συγκρίνουμε τις χώρες μεταξύ τους γιατί δεν υπάρχει καμία συνέπεια στη μεθοδολογία μεταξύ των διαφόρων κρατών και την ε, περιγραφή της πρόοδου. Και πέρα από αυτό βεβαίως δεν υπάρχει και πίνακας είπαμε όπου μπορεί κανείς να δει και να συγκρίνει στις διάφορες εκθέσεις χώρα τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει ούτε καν συγκριτικός πίνακας ε, των περισσινών συστάσεων για την ίδια χώρα σε σχέση με τις φετινές για να μπορούν πιο εύκολα οι δημοσιογράφοι να καταλαβαίνουν το κοινό τι γίνεται ότι τα θεσμικά όργανα εργάζονται και για το κοινό και για τους ψηφοφόρους και ε, χρειάζεται να έχουμε αυτά, ε, αυτή την κριτική αξιολόγηση, εκτίμηση Πέρσι προέβημε σε κάποιες συστάσεις αποφάσεις στο Συμβούλιο πώς υλοποιήθηκαν υπάρχει εύκολο τρόπο να το συγκρίνετε. Αν δεν το κάνετε αυτό, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν κάνετε καλά τη δουλειά σα. Και θολώνετε και τα νερά. Εντάξει, ε, η κυρία Φερέιρα τώρα. Για 10 λεπτά μέχρι τη λέξη της συνεδρίασης. Ευχαριστώ, αλλά δεν χρειάζομαι 10 λεπτά. Ναι, για να προσπαθήσω να αντιδράσω στις παρεμβάσεις θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας του συναδέλφους για τις προτάσεις του και θα ήθελα κυρίως να τους ευχαριστήσω για τις βελτιώσεις που πρότειναν ε, και που θα ε, βελτιώσουν την έκθεση σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Γκοζέσα σύμφωνα πλήρως με την ερμηνεία του. Είναι κάτι που το Κοινοβούλιο κάνει, που το Κοινοβούλιο ζητάει πάντοτε να γίνει αυτό και εκείνο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν να μην συνέβαινε τίποτα και νομίζω ότι εάν έχουμε ένα κονσένσους, γευρημένο κονσένσους σχετικά με ορισμένες συστάσεις, θα έπρεπε να περάσουμε σε μια πιο εντατική φάση, ούτως ώστε να υλοποιηθούν πραγματικά οι πρωτοβουλίες, να γίνουν και πιο συγκεκριμένες, διότι οι πολίτες ε, είναι, βρίσκονται σε απόγνωση σε ορισμένες χώρες. Δεν καταλαβαίνουν ε, ε, ποιος οδηγεί αυτό το μεγάλο όχημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ που ρωτήσατε τον Μάριο Ντράγκη πώς ερμήνευε την κατάσταση στην Πορτογαλία. Όχι επειδή είναι η χώρα μου, αλλά επειδή απλώς είναι μια χώρα που μέχρι τα όρια ακολούθησε όλες τις συστάσεις της Τρόικα και όμως δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Ε, ο Υπουργός έδωσε την παρέτησή του, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, απόγνωση και κανείς στην Τρόικα δεν προσπαθεί να αξιολογήσει τις συστάσεις που έγιναν στις χώρες. Ένα μήνυμο ανάλυση για να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Αυτό είναι το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς να κάνει όταν ε, η εμπιστοσύνη κλονίζεται. Ε, πρέπει να γίνει μια ανάλυση, μια ανάλυση παράλληλα με αυτή που ζήτησε ο Γκίγκολ. Ο Γκίγκολ ζήτησε να κάνουμε, να γίνει μια ανάλυση των ε, προγενέστερων συστάσεων. Εγώ συμφωνώ, συμφωνώ πλήρως, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό οι συστάσεις ακολουθήθηκαν. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια διαφορετική ανάλυση για την ποιότητα των συστάσεων. Γιατί μια χώρα που ακολουθεί τυφλά αυτές τις συστάσεις καταλήγει σε μια κατάσταση σοβαρότερη από αυτήν που θα είχε αν δεν είχε ακολουθήσει τις συστάσεις. Αυτό απαιτεί ενδελεχή ανάλυση πρέπει να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα, να δούμε τι έχει γίνει και αν είναι απαραίτητο ίσως να αναθεωρήσουμε ε, τις ε, τα διάφορα στάδια της διαδρομής όσον αφορά τα άλλα σχόλια. Δεν εκπλήσουμε που ο κύριος Έπινγκ ε, ανέφερε ορισμένα προβλήματα που γνωρίζω καλά είναι κατά του ΣΕΣΕΗ, κατά του κοινωνικού πυλώνα και του γεγονότος ότι οι μισθοί ε, ευθυγραμμίζονται με την, ε, με την ανταγωνιστικότητα. Αλλά όταν υπάρχει μείωση της ανταγωνιστικότητας, τι γίνεται και αυτό που είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί και εξάλλου το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν κάνει ορισμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Το Κοινοβούλιο ήδη έχει λάβει θέση ε, σχετικά με τον φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, για τον κοινωνικό πυλώνα και για την ΣΕΣΕΗ. Περιμένουμε την πρόταση. Καταλαβαίνω ε, την άποψή του, αλλά δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα όσα είπε ο Φίλιπ Λομπέρ. Συμφωνώ με ορισμένες από αυτές τις παρατηρήσεις και ελπίζω ότι ορισμένες από αυτές θα φτάσουν σε άλλα επίπεδα γενικής συνένεσης, κονσένσους. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει μια σύγκληση σχετικά με την γενική γραμμή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, περιμένω απλώς τις τροπολογίες για την έκθεση αυτή, αλλά θα ήθελα ειλικρινά, όπως το είπε ο κύριος Γκοζές, να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, να συγκεκριμενοποιήσουμε την ημερήσια διάταξη, να υπάρχει περισσότερη πίεση από αυτό το κοινοβούλιο για να απαντήσουμε στο άγχος ε, των πολιτών που βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της έλλειψης προσανατολισμού στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Thank Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Φερέιρα. Δυστυχώς, λόγω του κατεπίγουσας ανάγκης αυτής της έκθεσης, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 17 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση για σήμερα. Θα επανέλθουμε στις 3 ε, το απόγευμα.